Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων καθώς και του ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα 2020. Με χαρά σας ενημερώνω ότι αριθμός ρεκόρ βουλευτών, δηλαδή 116 βουλευτές από τα 27 Εθνικά Κοινοβούλια της Ένωσης, δύο μέλη από τις υποψήφιες χώρες και ένας μέλος από τις χώρες παρατηρητές έχουν εγγραφεί για την φετινή εκδήλωση. Αυτή η κοινοβουλευτική διάσκεψη εστιάζει στη διεύρυνση και εμβάθυνση της οικονομικής και τη διακυβέρνηση μάλλον τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θα ήθελα να σα πω δύο λόγια από την άποψη, την πλευρά μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το, Euro είναι, το ευρώ είναι ένα από τα πιο ορατά σύμβολα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και είμαστε ευχαριστημένοι που πάνω από, τους, από ένα στου τρει Ευρωπαίου πολίτε θεωρούν ότι το ενιαίο νόμισμα είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση υψηλότερη υποστήριξη που έχουμε δει από την εισαγωγή του ευρώ το 2002. Ελπίζουμε πως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορέσουν να ωφεληθούν από το ευρώ και καλωσορίζουμε την πρόθεση της Κροατίας και της Βουλγαρίας να να ε, δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να μπουν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ισοτιμιών. Πέρα από όλα αυτά θα πρέπει να μιλήσουμε όμως και για τις ευάλωτες πλευρές του κοινού μας νομίσματος που εκτέθηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντική πρόοδο στην ολοκλήρωση της ΟΝΕ, ε, ναι. κάποια μειονεκτήματα και διαρθρωτικά προβλήματα που ήταν αντικείμενα πολυάριθμων ψηφισμάτων του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ, τη οποία προεδρεύω, θα συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προχωρήσουμε στο πλαίσιο εκθέσεων ίδια πρωτοβουλία για την περαιτέρω ανάπτυξη τη ε, Ένωση Κεφαλαγορών, την αναθεώρηση του μακροοικονομικού νομοθετικού πλαισίου για καλύτερο αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία τη Ευρώπη και τη βελτιωμένη ε, διαφάνεια στην ε, λήψη αποφάσεων και το δημοκρατικό έλεγχο, ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και τέλος σε ψηφιακή οικονομία, αναδυόμενη κίνδυνη όσον αφορά τις κρυπτο... Ε, τα, τις κρυπτο ε, τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία. Επίσης συνεχίζουμε να εξετάζουμε το, πρόβλημα, το πρόγραμμα EDIS ε, που είναι ο πυλώνα που λείπει από την Τραπεζική Ένωση και ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε τα, ε, στο πρόγραμμα, στις προθέσεις του Συμβουλίου το πρόγραμμα δημοσιονομικού μέσου για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Στο τέλος του χρόνου αναμένουμε από την Κομισιό πρόταση για το ε, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ε, Αντασφάλισης για την Ανεργία που στόχο έχει να βοηθήσει εκείνους που έχουν μείνει χωρίς δουλειά λόγω εξωτερικών σοκ. Τέλος, ε, σε αρκετές, με αρκετές ευκαιρίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει για την ενίσχυση της του δημοκρατικού ελέγχου και θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων για το πώς ο ρόλος τους θα μπορούσε να ενισχυθεί στον έλεγχο των αποφάσεων των εθνικών τους κυβερνήσεων όσον αφορά τα θέματα της ΟΝΕ. Πριν δώσω το λόγο στους συγκεκριμένους προσκεκλημένους μας, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποιους κανόνες για τη διεξαγωγή αυτής της συνέλευσης. Επειδή είναι μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων, παρακαλώ να κατανοήσετε ότι μετά από τις εισαγωγικές παρατηρήσεις των καλεσμένων μας, μάλλον δεν θα είναι δυνατόν όλοι να πάρετε το λόγο σήμερα ε, και γι' αυτό το λόγο σας ζητώ να κρατήσετε τις παρεμβάσεις στο δίλεπτο ή τρίλεπτο το πολύ, όπου θα βλέπετε στο ε, ρολόι που θα αναγράφεται στον πίνακα. Αυτό ισχύει και για τους ευρωβουλευτές και για τους ε, εθνικούς βουλευτές. Θα έχετε δε κάποιες κάρτες ομιλίας με τις οποίες μπορείτε να υποδείξετε πως επιθυμείτε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν να συμπληρώνετε τις κάρτες αυτές και να τις δίνετε στους κλητήρες. Αυτό ισχύει όπως είπαμε και για τους ε, εθνικούς βουλευτές και για τους ευρωβουλευτές. Εν γέννη προσπαθούμε να μοιράσουμε το χρόνο ομιλίας ως εξή Δύο εθνικοί βουλευτές, ένας ευρωβουλευτής και ούτω καθεξής. Και πάλι, εάν υπάρξει ανάγκη, θα προσαρμόσουμε ίσως αυτή τη μέθοδο στη διάρκεια της συζήτηση. Θα δούμε δηλαδή πώς θα πάνε τα πράγματα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Κροσδάνα Πέριτς, που είναι πρόεδρος ε, του Επιτροπή Οικονομίας και προπολογισμού του Κρατικού Κοινοβουλίου. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω κρατικά, οπότε παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε κοντά μας τον Προεδρεύοντα του ΕΚΟΦΗΝ και ε, ε, Υπουργό Οικονομικών της Κροατίας, τον κύριο Μάριο Σεντένο, πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Βάλτης ε, Ντομπρόφσκης, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τζεντιλόνι, που είναι επίτροπος αρμόδιος για την οικονομία Αγαπητοί ε, εθνικοί βουλευτές και αγαπητοί ευρωβουλευτές, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Περιφερειών και της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η Κροατική Προεδρία είναι μια ιστορική στιγμή για μας. 28 χρόνια μετά την ε, ανεξαρτησία της Κροατίας, Ακολουθήσαμε την ε, προενταξιακή διαδικασία και την ενταξιακή διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την ένταξη της χώρας μας τον Ιούλιο του 2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφτά χρόνια λοιπόν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που προεδρεύουμε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξεκινάμε ένα νέο κύκλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κροατία είναι ένα σχέδιο ειρήνης άνευ προηγουμένου. Πρόκειται για μια μια κοινότητα που βασίζεται στην αλληλεγγύη και τις κοινέ αξίες. Η κρατική Προεδρία φτάνει σε μια στιγμή κλειδί και έχουμε έτσι την ευκαιρία ως κρατία να δώσουμε μια νέα όθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε τη διαδικασία εκδημοκρατισμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τρόπο ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε αυτό που αναμένουν οι πολίτες από εμά. Το σύνθημά μας είναι μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Αυτό που έχει σημασία στην Ευρώπη είναι οι αξίες και θέλουμε να τις ενισχύσουμε και να απαντήσουμε σε όλες τις σημερινές προκλήσεις. Με ιδιαίτερη χαρά εκφράζομαι στο όνομα των, ε, βουλευτών της Κροατίας και χαίρομαι που συμπροεδρεύω με την κυρία ε, την άλλη που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ του Ευρωκοινοβουλίου. Το ευρώ έχει ενισχυθεί την τελευταία δεκαετία και αυτό χάρη σε μια χρηστή οικονομική διακυβέρνηση και εμείς θα συνεχίσουμε να συζητάμε στα διάφορα επίπεδα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω το ευρώ και περιμένω με ανυπομονησία τις σημερινές μας ε, συζητήσεις. Και τώρα, χωρίς να καθυστερήσω άλλο, θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Μάρης, πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ, για να μας μιλήσει για τις προτεραιότητες του ΕΚΟΦΗΝ. Παρακαλώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κυρία Τινιάλη, κυρία Πέριτ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, πρόεδρε του Eurogroup, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη Κομισιόν, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να καλούμε να συμμετάσχω σε αυτή τη διάσκεψη που η Κροατία έχει την τιμή να οργανώσει φέτο μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ανταλλαγέ μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικέ για τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Και είναι πράγματι η κατάλληλη στιγμή να δούμε εκ το σύνεγγυ το πλαίσιο τη οικονομική διακυβέρνηση. Ένα λόγο είναι ότι ξεκινάμε ένα νέο θεσμικό κύκλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πάντοτε αποτελεί μια καλή ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα προ τα πίσω και να θεωρήσουμε τι έχουμε ήδη πετύχει και που θέλουμε να Πάμε στη συνέχεια. Ένα άλλο καλό λόγο είναι ότι οι περισσότεροι κανόνε οικονομική διακυβέρνηση θεσπίστηκαν περίπου πριν μια δεκαετία, απαντώντα ε, στην παγκόσμια κρίση χρέους ε, και από αυτή την ε, οπτική τώρα μπορούμε να δούμε πίσω και να δηλώσουμε ότι πολλά έχουν επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία δεκαέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε τους κανόνες για το συντονισμό πολιτικής ε, πιο πολύπλοκους και τους επέκτηνε πέρα από τις δημοσιονομικές πολιτικές. Επίσης δημιουργήθηκε και ο μηχανισμός Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα για να δοθεί μία απάντηση στι σοβαρέ απειλέ τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Επίση, έχει δημιουργήσει την Τραπεζική Ένωση που έχει τώρα το Μηχανισμό Εξηγήσεω Τραπεζών και το Μηχανισμό Εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εισαγάγει νέα μέσα νομισματική πολιτική. Όλε αυτέ οι βελτιώσει έχουν κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη πιο ισχυρή, έχοντα καλύτερα μέσα για να μετωπίσει τι υφέσει από ό,τι πριν μια δεκαετία. Οι νέοι κανόνε έδωσαν κίνητρα στα κράτη-μέλη για να μειώσουν ε, κάποιε ανισορροπίε που είχαν συσσωρεύσει στο παρελθόν. Όμω, βάσει πρόσφατη ανάλυση, οι νέοι κανόνε δεν είχαν αντίκτυπο στην προκυκλικότητα των δημοσιονομικών πολιτικών και ε, η εποχή ε, τη καλή οικονομία δεν χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθούν δημοσιονομικά μαξιλάρια ασφαλεία. Όμω πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτοί οι κανόνε είχαν ε, σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Τότε, σήμερα, αντιμετωπίσουμε διαφορετικέ προκλήσει. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλό πληθυσμό και χαμηλά επιτόκια. Θα πρέπει να βρούμε τρόπου για να εναγκαλίσουμε την τεχνολογία που εξελίσσεται και την καινοτομία με τι κοινωνικέ και οικονομικέ συνέπειέ του. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και ιδίω δημογραφικά ζητήματα που είναι ολοένα και πιο πολύπλοκά, κυρίω σε κάποια από τα νεότερα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε του κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι οικονομίε μα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με το εμπόριο. Πρέπει να σκεφτούμε για το μέλλον και να διασφαλίσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει εύρωστη και σε αυτό το και ευημερεί σε αυτό το περιβάλλον που εντελώ, συνεχώς αλλάζει. Συζητήσεις ε, για πιθανές βελτιώσεις ε, στο πλαίσιο κυβέρνηση είναι απαραίτητε για να απαντήσουμε τις νέες ε, ανάγκες και προκλήσεις. Ενώ προωθούμε οικονομική σταθερότητα και η φόρο ανάπτυξη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Η Κομισιόν πρόσφατα έκανε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή με την ανακοίνωσή τη για την αναθεώρηση τη διακυβέρνηση. Η ανακοίνωση μα δίνει μια καλή ανάλυση τη αποτελεσματικότητα της, ε, του σημερινού πλαισίου οικονομική διακυβέρνηση και θέτει τα σωστά ερωτήματα. Επίση, ανυπομονώ να δω τα αποτελέσματα τη δημοσίας διαβούλευση αυτής της ανασκόπηση που ξεκίνησε χτε. Είμαι βέβαιο ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εθνικέ αρχέ και τα κοινοβούλια θα συνεισφέρουν ενεργά στη συζήτηση αυτή. Ως ε, Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια ανταλλαγή ε, απόψεων ε, για το 2-pack και το 6-pack ε, στην ε, άτυπη συνάντηση Υπουργών Οικονομικών που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο στο Ζάγκρεπ. Εκεί θα επικεντρωθούμε στην διαδικασία μακροοικονομικών ενισορροπιών. Σήμερα στη συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ, σήμερα το πρωί, ακούσαμε την παρουσίαση τη Κομισιόν για την αναθεώρηση του πλαισίου διακυβέρνηση. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τομεί όπου οι απόψει των κρατών μελών θα συγκλίνουν. Οι περισσότεροι από εμά θα συμφωνούσαν ότι τα δημοσιονομικά πλαίσια θα πρέπει να προωθήσουν τι επενδύσει κυρίω σε μια πράσινη και ψηφιακή οικονομία και, η μετάβαση προς, και τη μετάβαση προ αυτή, ενώ θα διασφαλίσουμε μικροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα. Γενικότερα, το να αυξήσουμε την ποιότητα ε, και την φιλική προστασία των δημοσίων οικονομικών θα πρέπει να την κατοπτρίζεται καλύτερα στη διακυβέρνησή μα. Πολλοί επίση θα συμφωνούσαν ότι πρέπει να προωθήσουμε την εθνική κυριότητα και επομένω θα πρέπει να έχουμε πιο απλού κανόνε που θα βασίζονται σε ε, οικονομικέ μεταβλητέ ε, που θα μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο. Είναι σημαντικό να έχουμε συντονισμό ε, που θα βασίζεται σε βελτιωμένο συντονισμό. Όμω πρέπει επίση να εμβαθύνουμε την πρόοδο για να εμβαθύνουμε την ΟΝΕΗ. Η Κροατία δεσμεύεται για σε αυτό το πρόγραμμα, όχι μόνο ω Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ε, επειδή θέλουμε να μπούμε σύντομα στην Ευρωζώνη, αλλά επειδή είμαστε και πεπισμένοι ότι μία ΟΝΕ που λειτουργεί καλά είναι προ το συμφέρον όλων των κρατών μελών. Το ευρώ είναι το νόμισμα τη Ένωση και τα περισσότερα κράτη-μέλη αναμένεται να το υθετήσουν κάποια στιγμή. επομένω, είναι σκόπιμο όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στη συζήτηση για την εμβάθυνση τη ΟΝΕ. Είμαι βεβαίω ότι ο Μάριο, πρόεδρος του Eurogroup, θα έχει πολλά να πει για αυτό το θέμα σήμερα, καθώ το Eurogroup εργάζεται στο θέμα τη εμβάθυνση ε, τη ΟΝΕ βάσει εντολή από του ηγέτε. Όμω να πω δύο λόγια για το τι πιστεύουμε εμεί ότι θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητε για το νομοθετικό θεματολόγιο στον τομέα αυτό ω Προεδρία. Ο πρώτο μας είναι να ολοκληρώσουμε τη θέση του Συμβουλίου για το δημοσιονομικό εργαλείο για τη σύγκληση και την αγωνιστικότητα για την Ευρωζώνη και τα ενδιαφέροντα μέλη που ανήκουν στο Μηχανισμό Συνολικματικών Ισοτιμιών 2. Ε, η λιπόφαση λήφθη το Δεκέμβριο του 2018. Η νομοθετική δουλειά βασίζεται στην πρόταση τη Κομισιόν για το πρόγραμμα στήριξη μεταρρυθμίσεων καθώ και το, ΣΥΤΕ για το, για το Term City για τον BIC που συμφωνήθηκε από το Eurogroup πέρσι τον Οκτώβριο. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτό το φάκελο. Το κοινό δημοσιονομικό μέσο που θα υποστηρίξει την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα ανταγωνιστικότητα είναι σημαντικό για χώρες ε, που έχουν ε, ενωπήσει την κυριαρχία τους σε σχέση με νομισματική πολιτική και σε σχέση με τα μέσα ανασυναλλαγματικών ισοτιμιών. Πιστεύω ότι και το Κοινοβούλιο δίνει μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τον τριμερή διάλογο αυτό το εξάμεινο. Ένα βασικό στοιχείο προς ε, μια ανεξάρτητη και ισχυρή ΟΝΕ είναι ένας τραπεζικός τομέας που θα μπορεί να διαχειρίζεται καλύτερα τη κρίση, θα έχει λιγότερους κινδύνους και θα επιμερίζεται τους κινδύνους. Δηλαδή, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και το κομμάτι ε, που λείπει, που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων. Έχει σημειωθεί πρόοδος για το σύστημα καταθέσεων, όμως είναι πολύπλοκο το θέμα. Το να πετύχουμε αυτό το θέμα θα χρειαστεί ε, χρονοβόρες συζητήσεις. Εμείς σκοπεύουμε να τις συνεχίσουμε σε στενή συνεργασία με την Προεδρία του Eurogroup. Υπό την Προεδρία μας, το Συμβούλιο θα συνεχίσει τις τεχνικές συζητήσεις για το σχεδιασμό του μελλοντικού ίντις. Επίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε στην δημοσιονομική ολοκλήρωση και θα πρέπει να έχουμε σημειώσουμε πρόοδο με την Ένωση Κελαφοράς. Οι κεφαλαγορέ στην Ευρώπη είναι πολύ κατακαιρματισμένες για να μπορέσουν να προσφέρουν πλήρη ωφέλου στους επενδυτέ στι επιχειρήσει και στι οικονομίε. Μια ισχυρή τραπεζική ένωση μαζί με μια πλήρη ένωση κεφαλαγορά είναι ο δρόμος για το ευρώ για να έχει έναν ισχυρότερο ρόλο διεθνώ. Και αυτή είναι μια από τι προτεραιότητε που θα συζητήσουμε στο Ζάγκρεπ, στο ΕΚΟΦΗΝ, κατά την Προεδρία μα. Ε, θέλουμε να καταβάλουμε προσπάθεια για να θέσουμε σε εφαρμογή και τα υπόλοιπα μέτρα για το αναφερμένο σχέδιο για να δημιουργήσουμε την Ένωση Κεφαλαγορών. Επίση, θα υποστηρίξουμε τον καθορισμό νέων προτεραιοτήτων ε, που ε, θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση του νέου σχεδίου δράση για τον επόμενο θεσμικό κύκλο. Όπω βλέπετε, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα. Είναι αλλά ένα και πιο σημαντική δεδομένου του διεθνού τοπίου στο οποίο βρίσκεται η Ευρώπη σήμερα ε, οι κανόνες ε, και ε, ο τρόπος συνεργασίας που να εδώ και καιρό αντιμετωπίζουν αμφισβήτηση τα προβλήματα της κοινωνίας και του περιβάλλοντος χρήζουν ριζοσπαστικών λύσεων για τις επόμενες γενιές. Πρέπει λοιπόν εδώ σε Ένωση να διασφαλίσουμε ότι κατανοούμε τις ανησυχίες ο ένας του άλλου και να εργαστούμε για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για όλους και για το μέλλον των πολιτών μας. Εγώ ε, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και ανυπομονώ για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Μάριτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάριτς. Ο επόμενος ομιλητή μα είναι ο Μάριος Σεντένο, πρόεδρος του Eurogroup. Θα μας συζητήσει, θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες του Eurogroup. Ευχαριστώ πολύ, συμπρόεδροι, εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της Κομισιόν. Είναι η τιμή μου που συμμετέχω σε αυτήν την ε, διάσκεψη στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας 2020. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω όπως και στη Λισαβόνα, στο δικό μου, στη δική μου χώρα. Έχω συμμετάσχει σε περίπου 30 κοινοβουλευτικέ συνελεύσει ετησίω Είναι σημαντική η πολιτική συζήτηση και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που βελτιώνουν τις πολιτικές και βελτιώνουν τη στιβαρότητα της δημοκρατίας μας. Θα σας μιλήσω για την διακυβέρνηση σε επίπεδο ευρωζώνης που είναι πιο περίπλοκη από τη σε εθνικό επίπεδο αλλά εξίσου σημαντική. Κυρίες και κύριοι, η στήριξη για το ενιαίο νόμισμα μεταξύ Ευρωπαίων είναι στο 75 περίπου της 100 σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο. Αυτό είναι το υψηλότερο νούμερο που πιάσαμε ποτέ. Ε, είμαστε περήφανοι Ευρωπαίοι που καταλαβαίνουμε την αξία του ευρώ. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους πολίτες μας. Ε, ε, δημιουργήσαμε πριν από 20 χρόνια περίπου το ευρώ, αλλά ακόμη δεν έχουμε στελεχώσει σωστά τα ε, θεσμικά όργανα. Η διακυβέρνηση πρέπει ακόμα να αναπτυχθεί. Αυτό είναι σημαντικό και ήταν κατά την κρίση. Από τότε κάναμε βήματα για να ολοκληρώσουμε θεσμικά ε, τη θέση μας. Σήμερα πρέπει να προστατέψουμε τους πολίτες, το νομισμά μας απέναντι σε κινδύνους και παγίδες. Πολλά έχουν γίνει, πολλά εξακολουθούν να γίνονται. Μετά ε, την κρίση ε, τώρα υπάρχει μια επιβράδυνση. Η συζήτηση για την, διακυβέρνηση της ΟΝΕ είναι επίκαιρο θέμα που χρειάζεται να γίνει. Η διακυβέρνηση της ΟΝΕ καλύπτει τρία πράγματα. Πρώτον, υπάρχουν κοινοί κανόνες που διέπουν τα δημοσιονομικά ε, και οικονομικά των κρατών μελών. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά της διακυβέρνησης. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο ίσως είναι το καλύτερο παράδειγμα εδώ. Γενικά είμαι πεπισμένος ότι το πλαίσιο των κανόνων μας ε, βοήθησε και εμάς και τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν συσσωρευμένες ανισορροπίες. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης εξαρτάται και τα θεσμικά όργανα. Τα κοινά θεσμικά όργανα που έχουμε δημιουργήσει έφεραν σε νέο επίπεδο τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ. Τρίτον, η διακυβέρνηση της ΟΝΕ εξαρτάται και από συζητήσεις, ε, πίεση των ομολόγων ε, και συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό δημιουργήθηκε και το Eurogroup μεταξύ άλλων και αυτός είναι ο ρόλος του με βάση τη συνθήκη της Ένωσης. Ο ρόλο του Eurogroup στην κρίση καταδεικνύει τη σημασία του. Επίσης, διαμορφώνουμε όλο και περισσότερο και δομούμε τις άτυπε διαδικασίες συντονισμού. Για παράδειγμα, για να δείξω αυτό που αναφέρεται ως ήπιος συντονισμό ε, είναι ο fiscal stance τους προηγούμενους μήνες. Το Eurogroup έκανε πολλές συζητήσεις για τις οικονομικές προοπτικές και το κατάλληλο μείγμα πολιτικής. Τώρα τα κράτη-μέλη καλούνται να ε, προσαρμόσουν τα δημοσιονομικά τους στον υφιστάμενο δημοσιονομικό χώρο. Η δημοσιονομική αντίδραση θα πρέπει να είναι ε, μια θέση πιο υποστηρικτική σε συνολικό επίπεδο, τηρώντας τους δημοσιονομικούς κανόνες. Γίνονται συστάσεις αναχώρα. Οι χώρες θα αξιολογούνται με βάση αυτό το πλαίσιο πολιτικής ο πολιτικός συντονισμός ή ο συντονισμός των πολιτικών σε ενωσιακό επίπεδο έτσι λειτουργεί. Είναι αποτελεσματικός. Αυτό είναι θεμητό ερώτημα. Η κρίση βοήθησε να εξυγχρονίσουμε τον επιχειρηματικό μας κύκλο και τώρα έχουμε την μικρότερη διασπορά ε, των δημοσιονομικών θέσεων. Υπάρχει χώρος και περιθώριο για βελτίωση, περαιτέρω ολοκλήρωση. Έτσι η νομισματική μας πολιτική θα καταστεί αποτελεσματικότερη. Όσοι ε, έχουν τα πράγματα η πρόοδος ε, βελτιώνει τη διακυβέρνηση γενικότερα. Ε, η Ευρωζώνη έγινε πιο ανθεκτική. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος σήμερα διαφέρει από την πριν από 10 χρόνια. Αντιμετωπίζουμε τις κλιματικές προκλήσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό που απαιτούν κατεπίγουσα και συλλογική δράση. Επίσης υπάρχουν γεωπολιτικές εντάσεις ε, Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες που σχετίζονται και με τις εμπορικές σχέσεις. Έχουμε να κάνουμε κρίσιμες επιλογές και αυτές είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αν θέλουμε να ε, κατοχυρώσουμε την οικονομική μας κυριαρχία. Πάνω σε αυτή τη βάση, καλό είναι ένα απολογισμό να δούμε αν η διακυβέρνηση τη ΟΝΕ εξακολουθεί να ανταποκρίνεται ε, στι ανάγκε. Εμεί χαιρετήσαμε την, την αναθεώρηση των κανόνων. Ε, το Eurogroup ε, θα αρχίσει τη διαδικασία διαβουλεύσεων που γίνεται σχετικά τα προηγούμενα δύο χρόνια. Επίσης ε, αναθεωρήσαμε την, ε, ε, ε, στην πολιτική μας σε θεσμικό επίπεδο. αυτό το έργο δεν ήταν μόνο τεχνικά περίπλοκο αλλά και πολιτικά ευαίσθητο απαιτούσε μακρές συζητήσεις και ισορροπημένες λύσεις. Να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση του έργου μας και τα επόμενα βήματα. Καταρχήν το νομισματικό εργαλείο για την Ευρωζώνη είναι το πιο καινούριο project για την εμβάθυνση. Προετοιμάσαμε την ε, συμφωνία του 2018 στο Συμβούλιο Κορυφής ε, και το 2019 το Eurogroup συζητήσαμε τις ε, αρχές που θα διέπουν το νέο αυτό εργαλείο. Ας δούμε ποια είναι τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Συμφωνήσαμε ότι το μέσον αυτό πρέπει να συγχρηματοδοτεί εθνικές μεταρρυθμίσεις και δημόσιες επενδύσεις με στόχο την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωζώνη. Η σύγκληση δεν είναι φυσικό αποτέλεσμα ε, της ε, νομισματικής ε, ολοκλήρωσης. Θέλει και εθνικές πολιτικές υπέρ των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων. Θέλει ειδικό προπολογισμό για τις χώρες της Ευρωζώνης. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις ε, επίσης θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικέ. Όσο πιο πολύ συγκλίνει και όσο πιο ανταγωνιστική είναι η Ευρωζώνη, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η νομισματική πολιτική της ε, Κεντρικής Τράπεζας και τόσο περισσότερους καρπούς θα δρέψουν οι πολίτες. Οι δημόσιες ε, επενδύσεις ε, θα πρέπει να συνεχίζονται στην κρίση. Ε, γι' αυτό έχουμε συγκριματοδότηση σε χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Επίσης προβλέπουμε ευέλικτο ε, επιμερισμό ε, κονδυλίων στις χώρες για να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες προκλήσεις. Τον Ιούνιο του 2019 η Σύνοδος Κορυφής υπογράμμισε την σημασία της λήψης αποφάσεων των κρατών μελών. Στρατηγικές αποφάσεις ε, που στηρίζονται από το ε, νέο μέσο θα ε, δίδονται από το Σύνοδο Κορυφής και το Eurogroup που θα συζητήσουν και άλλες προτάσεις χωρών για να αντιμετωπιστούν χρηματοδοτικά νέες ανάγκες ο συντονισμός των πολιτικών θα πρέπει να ενισχυθεί και θα πρέπει οι ευρωπαϊκές πολιτικές να εφαρμόζονται, να ε, θεωρούνται δικές δικές μας πολιτικές, πολιτικές των κρατών μελών. Η εφαρμογή του δημοσιονομικού μέσου θα ε, υπόκειται στον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Ευρωκοινοβουλίου. Υπολογίζω στην υποστήριξή σας, ε, στην βοήθειά σας. Τα εθνικά κοινοβούλια προφανώς μπορεί να παίξουν και εκείνα ρόλο, ε, προετοιμάζοντας τις προτάσεις των χωρών για την Σύνοδο Κορυφής. Ε, τώρα, κάποια δημοσιονομικά στοιχεία. Οι ηγέτες αποφάσισαν ότι το μέσον θα είναι μέρος του ενωσιακού προϋπολογισμού ε, και θα αποφασίζεται από τους ηγέτες. Δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα των συζητήσεών τους, είναι πιθανόν όμως το μέγεθος του μέσου αυτού, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, να είναι κάπως ε, μετριοπαθές. Ε, αυτή είναι πολιτική συζήτηση. Πιστεύω όμως ότι οι ηγέτε μας θα μπορέσουν να ενισχύσουν τη δύναμη πυρό του. Συζητήθηκαν οι πιθανέ δημοσιονομικές ε, χρηματοδοτικές πηγές του μέσου αυτού ε, θα μπορούσαν να διασφαλιστούν με χωριστή διακυβερνητική συμφωνία που είναι γνωστή ως IGA. Το Eurogroup συμφώνησε με μια έκθεση που παρουσιάζει τα θέματα που θα εξετάσουμε όταν φτάσουμε στο IGA. Η έκθεση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στους ηγέτες να ε, αποφασίσουν με πλήρη γνώση των θεμάτων. Τα 18 μέλη του Ευρωζώνης θα μπορέσουν έτσι να ε, αυξήσουν τον δημοσιονομικό φάκελο. Έχουμε ε, ευελιξία ο ενώ ενωσιακός προϋπολογισμός αναθεωρείται κάθε 7 χρόνια, εμεί κάθε έτος θέτουμε προτεραιότητες και πάντοτε ε, αντιμετωπίζουμε το ερώτημα έχουμε αρκετά, αρκετούς πόρους για να καλύψουμε τις ανάγκες αν η απάντηση είναι όχι θα πρέπει να αυξήσουμε τους πόρους του μέσου αυτού γι' αυτό οι συστάσεις της Ευρωζώνης είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι τόσο σημαντικές η διαφορά δεν είναι το μέγεθος αλλά η αποτελεσματικότητα θα έλεγα λοιπόν ότι η χρηματοδότηση του μέσου δεν είναι το, αυτό που μετράει πιο πολύ από όλα τώρα η πολιτική ε, σκοπό έχει να βρει μια σταθερά μεταξύ ρεαλισμού και μια ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και φιλοδοξίας στις επόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέσον θα ολοκληρωθούν όπως ελπίζω σύντομα ούτω ώστε το 2001 να καταστεί ε, λειτουργικό. Δύο λόγια τέλος ε, για κάποια άλλα ε, καθήκοντα της ΟΝΕ που απασχόλησαν πέρσι το Eurogroup. Πέρσι ε, καταλήξαμε σε σχέση με την αναθεωρημένη ε, συνθήκη και την ε, σχετική τεκμηρίωση. Θα ολοκληρώσουμε την πολιτική συζήτηση για την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να επικυρώσουν. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τα μέσα του 2021. Η αναθεώρηση της συνθήκης το, τα, θα τα κάνει πιο προσπελάσιμα, πιο προσβατά τα μέσα ε, προφύλαξης. Ε, όπως και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την πρόληψη κρίσεων στην Ευρωζώνη. Ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα είναι μια συμφωνία ότι το ESM θα πρέπει να έχει backstop για το ε, Ταμείο εξυγίανσης. Ε, κάνουμε τις απαραίτητες διευθετήσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως το 2021, τρία χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρόνο. Ε, τώρα, τρίτος πυλώνας ε, η ε, Τραπεζική Ένωση και η προστασία των καταθέσεων. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια πιο συνεκτική προσέγγιση. Πιο ολοκληρωμένος τραπεζικός τομέας για να μειώνονται οι κίνδυνοι, καλύτερη διαχείριση των κρίσεων και διασφαλίσεις για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτά γίνονται ε, στα, ε, υπό, την, υπό την ηγεσία του Eurogroup από τους ε, υφυπουργούς οικονομικών. Ε, όλοι κατάλαβαν τον κατεπήγοντα χαρακτήρα του θέματος. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε ένα πρόγραμμα δράσης ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την εντολή μας. Κοινή μας φιλοδοξία πρέπει να είναι να έχουμε πιο ολοκληρωμένη, πληρέστερη τραπεζική ένωση που θα γίνει μέχρι το τέλος της θητείας μας. Επίσης θα έχουμε κεφαλαία αγορές που ε, θα ε, παίξουν ε, βασικό ρόλο για την δημοσιονομική κυριαρχία της Ένωσης. Για να κλείσω, σημαντικές βελτιώσεις έγιναν μετά την κρίση για την διακυβέρνηση της ΟΝΕ. Έγινε πιο ανθεκτική η Ευρωζώνη. Το ευρώ βοήθησε να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της κρίσης. Έδρασε ως ασπίδα. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι σήμερα και οι πολίτες και οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές, οι ξένοι επενδυτές. Νέες προκλήσεις όμως ε, προέκυψαν. Έτσι είναι αναγκαία ε, μια αναθεώρηση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Ε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει, συνεχίζονται τα έργα για την εμβάθυνση της ε, ΟΝΕ. Η πολιτική βούληση έτσι αποδεικνύεται ότι υφίσταται. θα προχωρήσουμε αν και σταδιακά. Το Eurogroup συνεχώς προωθούσε τις αλλαγές και στις πολιτικές μας και θα συνεχίσει και στο μέλλον να παίζει το ρόλο του. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσω τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σεντένο. Μιλήσατε λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βάλτης Ντομπρόφσκης, αντιπρόεδρος της Κομισιόν, που θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές και ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ και υποστηρίζω την βαθύτερη και την πιο αποτελεσματική οικονομική και νομισματική ένωση. Ε, ε, είμαστε μέσα στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Πρέπει να προστατεύσουμε την ευημερία και τη σταθερότητά μας και να βοηθήσουμε τους ε, πολίτες και τις εταιρείε μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και πρέπει να ενισχύσουμε τη διεθνή μας αρχιτεκτονική. Η ισχυρότερη οικονομική και νομισματική ένωση απαιτεί ισχυρότερη διακυβέρνηση. Η πρόεδρος Βαντελάιεν κατέστησε σαφές στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές ότι η οικονομική διακυβέρνηση και δημοκρατικός έλεγχος ε, πηγαίνουν χέρι με χέρι. Ένα από τα διδάγματα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, ε, είναι ότι η συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων δημιουργούν περισσότερη αίσθηση οικειότητας με την Ευρωπαϊκή Ατζέντα και γι' αυτό και στόχος είναι να επισκεπτόμαστε τακτικά τα Εθνικά Κοινοβούλια για να ακούμε τις προτεραιότητές σας και να κερδίζουμε την υποστήριξή σας ώστε η φιλόδοξή μας ατζέντα να γίνει πραγματικότητα έχουμε τρία βασικά στοιχεία όπου ε, οφείλουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειες. Πρώτον, να επιταχύνουμε την πρόοδο όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση. Αυτό το project αφορά πρώτα απ' όλα την διασφάλιση των χρημάτων των φορολογούμενων, ώστε να μην πληρώνουν εκείνοι για τα σφάλματα των τραπεζών. Ταυτόχρονα χρειάζεται ισχυρό και ολοκληρωμένο δημοσιονομικό τομέα για να εξασφαλίσει τόσο η ε, δημοσιονομική μετάβαση όσο και η οι στόχοι της βιομηχανικής πολιτικής. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να ε, αναμέξει το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια στα θέματα και στις συζητήσεις για την Τραπεζική Ένωση, όπως είναι το πρόγραμμα εγγύησης καταθέσεων και το, πρόγραμμα, το Ταμείο Εξυγίανσης. Ε, ε, αυτά τα θέματα φαίνονται επίμαχα σήμερα, αλλά πρέπει να επιληθούν σήμερα για χάρη του κοινού μας μέλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τον αναθεωρούμε. Ελπίζουμε σύντομα θα ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια έτσι ώστε να έχουμε ενισχυμένο η εργαλειοθήκη ε, για μέτρα προληπτικά και ε, να ενταχθεί αυτό μέσα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης. Πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση, πράγμα που είναι όλο είναι και πιο σημαντικό από τη στιγμή που το, Ευρω... το Ηνωμένο Βασίλειο ε, βγήκε από την Ένωση. Υπάρχει συνένεση ότι χρειάζεται πιο βαθιά πιο βαθιές κεφαλαγορές και πιο ολοκληρωμένες κεφαλαγορές ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε και να δημιουργήσουμε και θέσεις απασχόλησης. Δεν είναι τεχνικά ο μόνο ζήτημα αλλά και πολύ ε, σημαντικό πολιτικής φύσης ε, θέμα γιατί ειδικά οι μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση ώστε να μπορέσουν να βαθμίσουν την Ευρώπη και γι' αυτό έχουμε και το Ταμείο για project ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Χρειάζεται επίση να δουλέψουμε περισσότερο για του επενδυτέ μικρή κλίμακα και να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στι κεφαλαίε γενικότερα. Πρέπει να προχωρήσουμε δε ε, γρηγορότερα ε, σε ένα, στο θέμα της ε, αφαιρεγκαιότητα και των διαδικασιών που αφορούν του τους φορολογικούς Καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει γίνει για το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα που θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των οικονομιών μας, κυρίως στις περιφέρειες, ε, δίνοντας κίνητρα για διαστατικές ε, ε, μεταρρυθμίσεις με οικονομική στήριξη. Επίσης εργαζόμαστε για το πρόγραμμα αντασφάλισης για τα επιδόματα τα ανεργία, ώστε να προστατευθούν οι πολίτε από εξωτερικά σοκ. Αυτό θα σημάνει περισσότερη συνοχή, σύγκληση μεταξύ των κρατών και θα ενισχύσει και την ΟΝΕ. Επιπλέον, αναθεώρηση της, του πλαισίου οικονομική διακυβέρνηση προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία ώστε να, να προχωρήσουμε σε ανοιχτέ συζητήσει για ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων για το πώ λειτουργούν οι κανόνε μα, πώ μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον. Ο Επίτροπο Τζεντιλόνι θα μιλήσει περισσότερο για αυτό το θέμα. Μία ζωντανή εύρωστη οικονομική ένωση βασίζεται στην ισοχρηστή οικονομική διακυβέρνηση, την τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαγορών έτσι ώστε να βελτιωθεί η οικονομική και ε, δημοσιονομική σταθερότητα της Ένωσης, να ενισχυθεί ο διεθνής ρόλος του ευρώ και να ενισχυθεί η οικονομική και δημοσιονομική μας αυτονομία. Επίσης αυτό θα ενισχύσει τη θέση μας και τη δράση μας στα διεθνή φόρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιπροσωπεύει ένα ανοιχτό και ε, μοντέλο που βασίζεται βασίζεται στην πολυμερή συνεργασία. Αυτό είναι και στόχος της Προέδρου για γεωπολιτικό κύρος της Ένωσης, διατήρηση και πρόθεση των αξιών μας και του μοντέλου ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Αυτός, ε, αυτό είναι το project μας και χρειαζόμαστε τους ευρωβουλευτές εσά και τους βουλευτές, εθνικούς βουλευτές για να δουλέψουμε πιο μια ισχυρότερη και πιο αποδοτική ΟΝΕ ναι, για ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντομπρόφσκης. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Παόλο Τζεντιλόνι, Επίτροπο Αρμόδιο για την Οικονομία ώστε να μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Τζεντιλόνι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που συμμετέχω αυτή την εβδομάδα, σε αυτή την κοινοβουλευτική εβδομάδα, η οποία αφιερώνεται στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό καθώς βρισκόμαστε σε μια στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνει τις αρμοδιότητές του και τα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι όλο ένα και πια επίκαιρα στην συζήτηση στο τελικό κοινοβούλιο. Και θα ήθελα τώρα να συνεχίσω στα αγγλικά. Λέγοντας ότι η συζήτηση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Καθώς, όπως υπενθύμισε ο Βάλτης, μόλις δημοσιεύτηκε η ανακοίνωση της Κομισιόν για την αναθεώρηση της οικονομικής διακυβέρνησης. Η συζήτηση λοιπόν για την οικονομική διακυβέρνηση έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Η οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ίσως είναι το πρώτο που πρέπει να αξιολογήσουμε στην ε, πρόσφατη χειμερινή μας πρόβλεψη. Ήταν ξεκάθαρο το μήνυμα σε σχέση με το ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη. Έχουμε σχεδόν 7 έτη ανάπτυξης, αλλά με ένα πολύ πιο βραδύ ρυθμό. Έτσι λοιπόν ε, κινδυνεύουμε να έχουμε χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλά επιτόκια, χαμηλό πληθωρισμό για μακρά περίοδο. Ταυτόχρονα έχουμε κάποιους εξωτερικούς κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση όπως παραδείγματος χάρη το ξέσπασμα του κορονοϊού στην Κίνα. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση, εξακολουθεί να υπάρχει ανάπτυξη, αλλά έχουμε και προκλήσεις ενώπιόν μας. Το δεύτερο σημείο είναι με την, έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα φιλόδοξε προκλήσει, συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ψηφιακή μετάβαση και το δημογραφικό. Όλα αυτά ε, ουσιαστικά αποτελούν ε, προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η Κομισιόν, αποστολές της Κομισιόν, αλλά και όλες αυτές οι αποστολές ε, σημαίνουν ότι είναι τεράστιες οι ανάγκες για επενδύσεις. Όμως ε, οι δημόσιες επενδύσεις εξακολουθούν κάτω από το επίπεδο πριν την κρίση. Η ανασκόπηση που ξεκινήσαμε πριν 10 χρόνια προσπαθεί να αξιολογήσει πώς λειτουργήσαν οι κανόνες μας την τελευταία δεκαετία, να στρέψει το βλέμμα της γύρω-γύρω και να δει σε ποιο πλαίσιο λειτουργούμε και να δει και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερους κανόνες. το να αξιολογήσουμε τι λειτουργήσε και τι όχι. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό. Σίγουρα μειώσαμε τα ελλείμματά μας και μετά από τη βαθιά κρίση είχαμε μία μικρά περίοδο ανάπτυξη. Επίσης μειώσαμε το χρέο μας, όμως ήταν διαφορετικό το επίπεδο της μείωσης σε διάφορες χώρες δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε προκλητικές πολιτικές και να μειώσουμε τα πλεονάσματα σε χώρες όπου υπήρχε δημοσιονομικός χώρος. Λεχθέν των αυτών για το παρελθόν, γενικά, οι κανόνες έφεραν καλά αποτελέσματα ως γενική εικόνα. Ταυτόχρονα όμως, στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε τους κανόνες αυτούς. Το ζήτημα δεν είναι να είμαστε υπέρ ή κατά εύρος των δημοσίων οικονομικών, αλλά έχει να κάνει με τη σύνθεση των δημοσίων οικονομικών. Το ζήτημα δεν έγκυται στο να καταργήσουμε τους κανόνες μας, αλλά να επικαιροποιήσουμε και να βελτιώσουμε τους κανόνες αυτούς για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Uh, Ποιοι είναι οι πιθανοί στόχοι των βελτιώσεων και της επικαιροποίηση, Θα ανέφερα δύο. δύο. Καταρχήν, να προσπαθήσουμε να πλουστεύσουμε τους κανόνες αυτούς. Είναι πολύ εύκολο στη θεωρία, αλλά όχι τόσο εύκολο στην πράξη. Γιατί συχνά η πολυπλοκότητα βοηθά την ευφυΐα. Είναι πολύπλοκοι λοιπόν οι κανόνες, γιατί πρέπει να έχεις και μία σειρά μέσων για να λάβεις τις σωστές αποφάσεις. Ταυτόχρονα όμως, αν η πολυπλοκότητα γίνει υπερβολική, γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκη λέει ο μιλητής, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή από τους πολίτες, από τους βουλευτές μας και από τις κυβερνήσεις μας. Και η διαφάνεια και η κυριότητα της διαδικασίας ε, τίθεται σε κίνδυνο. Ο δεύτερος στόχος είναι οι κανόνες αυτές, ε, αυτοί να είναι πιο φιλικοί προς την ανάπτυξη. Να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε τις επενδύσεις ε, που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ενωπιών μας. Νομίζω ότι μπορούμε να γεφυρώσουμε τις διαφωνίες μας, δεν είναι εύκολο, το γνωρίζω. Αλλά μπορούμε να γεφυρώσουμε τις διαφωνίες μας στη συζήτηση αυτή αν στρέψουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον και αν χρησιμοποιήσουμε την πολιτική μας βούληση. Και φυσικά έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση. Η συνεισφορά των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτή την ανοιχτή συζήτηση είναι ορθο τρόπο για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζεντιλόνη. Και τελευταίος ομιλητή είναι ο κύριο Φάμπιο Πανέτα, ο οποίο είναι μέλο του Εκτελεστικού Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα του δώσω το λόγο για να μιλήσει για την νομισματική πολιτική. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Επίτροπε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να λάβω το λόγο εδώ σήμερα. Η ΟΝΕ καλεί για συγχρονισμένες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που με τη σειρά τους απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και ημών, δηλαδή των Ευρωβουλευτών και των Εθνικών Βουλευτών. Ευθύ εξ αρχή, το εγχείρημα της ΟΝΕ συνοδεύτηκε από δύο κεντρικές συζητήσεις. Η πρώτη αφορά το τη σειρά της ολοκλήρωσης και το μέγεθος της ολοκλήρωσης. Κάποιοι έλεγαν ότι η πολιτική σύγκληση θα πρέπει να προηγηθεί τη νομισματική Ένωση, άλλοι έλεγαν ότι η οικονομική ολοκλήρωση θα προωθήσει την πολιτική ολοκλήρωση. Η δεύτερη συζήτηση αφορά το θέμα αν ε, ήδη ενσωματώνουμε νέα μέλη στην Ευρωζώνη ή θα πρέπει πρώτα να εμβαθύνουμε την θεσμική του ε, θωράκιση. Αυτές οι συζητήσεις ε, αναδεικνύουν επιλογές που πάνε πέρα από τις οικονομικές σκέψεις. Αντικατοπτρίζουν την κοινή βούληση της Ευρώπης να ε, συνενωθεί διαχρονικά. Η πολιτική αυτή δέσμευση απεδείχθη ισχυρότερη από ό,τι πίστευαν πολλοί. Αν όμως αυτή η δέσμευση πρόκειται να είναι ανθεκτική, θα πρέπει να υποστηρίζεται από αποτελεσματικές πολιτικές. Δύο προτεραιότητες βλέπω εγώ καθώς διευρύνεται η Ευρωζώνη η ανάγκη να γίνει η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ κατάλληλη για το σκοπό της ε, είναι ένα ζήτημα κατεπήγων. Δεύτερον, προς το συμφέρον των νέων και των υφισταμένων μέλων της Ευρωζώνης θα πρέπει συλλογικά να διασφαλίσουμε ότι ε, προετοιμάζεται σωστά η προσχώρηση, η διεύρυνση. Έτσι ε, δεν θα εμβαθύνει, δεν θα διευρυνθεί η ΟΝΕ πολύ γρήγορα. Τώρα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη της οικονομικής ολοκλήρωσης. Ε, αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντικό. Από μόνες τους οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι πολύ μικρές για να αντιμετωπίσουν παρεπόμενα από, και, ε, ε, από μεγάλες οικονομικές περιοχές, να έχουν μόχλευση στο διεθνές εμπόριο και στις σχετικές διαπραγματεύσεις ή να έχουν έναν σημαντικό διεθνή ρόλο για το νομισμά τους. Η συνεργασία λοιπόν είναι σημαντική. Η οικονομική ολοκλήρωση θα πρέπει να να τύχει αποτελεσματικής διαχείρισης αν θέλουμε να δρέψουμε πλήρη ωφέλη. Καθώς όλο και περισσότερες χώρες ε, εισέρχονται στην Ευρωζώνη, η οικονομική της δομή γίνεται πιο ε, διαφορετική και το ενδεχόμενο ε, παρεπόμενων ε, επιπτώσεων μεταξύ χωρών και δημοσιονομικών δομών γίνεται μεγαλύτερο. Αν ε, δεν είναι αποτελεσματική η διαχείριση, τότε η διασύνδεση μπορεί να επιβραδύνει την ΟΝΕ. Ε, κατά την κρίση η θεωρητική παρατήρηση έγινε πάρα πολύ πραγματική. Η ατελής φύση της ΩΝΕ οδήγησε σε μια ύφεση το 2012 και 2013 λόγω του χρέους που ήταν άνευ στην οικονομία της Ευρωζώνης. Η ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιμετώπισε την πρόκληση, αντιμετώπισε ε, την εντολή της, σταθεροποίησε τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στήριξε την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, δημιουργία θέσεων εργασίας. Μετά την αρχή της ανάκαμψης το 2013 η, οικονομία της Ευρωζώνης δημιούργησε πάνω από 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Σημαντικά βήματα πήραμε ώστε να γίνει πιο ανθεκτική η αρχιεκτονική της ε, ΟΝΕ, δημιουργώντας ε, κοινή τραπεζική εποπτεία, κοινό σύστημα να αντιμετωπίσει τις προβληματικές τράπεζες και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να βοηθήσει τις χώρες που είχαν ανάγκη. Όπως βλέπουμε όμως από τις πρόσφατες εξελίξεις, πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Ο πληθωρισμός είναι κάτω από το στόχο του ε, Συμβουλίου η ανάπτυξη δείχνει κάποια σημάδια σταθεροποίησης αλλά παραμένει ε, μικρή. Ε, πάνω σε αυτή τη βάση η οικονομία της Ευρωζώνης θα συνεχίσει να χρειάζεται υποστήριξη από την νομισματική μας πολιτική όσο χρειάζεται για να διασφαλίσουμε την ε, στιβαρή σύγκληση του πληθωρισμού προς το στόχο μας. Η ατελής φύση της ΟΝΕ είναι ένα κομμάτι αυτής της υπόθεσης. Η νομισματική πολιτική δεν υποστηρίχθηκε ε, επαρκώς από την ε, δημοσιονομική και άλλες πολιτικές και τη φορολογική πολιτική. Αυτό οδήγησε σε χαμηλότερη ανάπτυξη και ε, πληθωρισμό από ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά. Η κρίση μας θύμισε και πάλι ε, κάτι πολύ θεμελιώδες. Καθώς πρόκειται να διευρυνθεί η Ευρωζώνη θα πρέπει να ενισχύσει τη θεσμική της δομή. Ε, το πιο κατεπήγον καθήκον που αντιμετωπίζουμε είναι να ολοκληρώσουμε την Ένωση Τραπεζική και των Κεφαλαίων Αγορών ε, έτσι αυξάνοντας την ιδιοκτησία διασυνοριακά των περιουσιακών στοιχείων, στοιχείων ενεργητικού και δημιουργώντας πιο ισορροπημένη δημοσιονομική δομή. Η διαφορά στην Ευρωζώνη θα πρέπει να γίνει δύναμη και όχι αδυναμία. Οι ε, ε, οικονομικές ε, επιχειρήσεις θα διαφοροποιούνται σε ευρύτερο πλαίσιο και επίσης η αγορά θα μπορέσει να απορροφήσει οικονομικά σοκ μειώνοντας την ανάγκη για δημόσιο χρήμα. Καθώς διευρύνεται η Ευρωζώνη και καθώς οι προτιμήσεις των κρατών μελών γίνονται πιο διαφοροποιημένες ίσως θα είναι μεγαλύτερη η πρόκληση να βρεθεί συμφωνία επί τέτοιων εγχειρημάτων. Ε, αυτό δεν έχει να κάνει με ε, διαφορές, αλλά μάλλον διαφορές στη λήψη αποφάσεων. Αυτό δείχνει ότι θα πρέπει να έχουμε στεναρά θεσμικά όργανα με ξεκάθαρη εντολή και πλήρη δημοκρατική στήριξη, ιδιαίτερα καθώς διευρύνεται η Ευρωζώνη. Ε, θα πρέπει να έχουμε ε, θεματολόγιο για τη διεύρυνση και θεματολόγιο για την ε, εμβάθυνση της ΩΝΕ. Η εμπειρία δείχνει ότι η θηλοθέτηση του ενιαίου του κοινού νομίσματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ευκαιρίες. Δεν πρέπει να τις χάσουμε. Η ιστορία δίνει παραδείγματα ε, χαμένων ευκαιριών. Ε, διασφαλίζοντας ότι η νέα Ευρωζώνη θα αντιμετωπίσει τις οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις για επιτυχή συμμετοχή ε, είναι πάρα πολύ σημαντική και εξυπηρετεί τους πάντες. Είναι πολύ σημαντικό οι χώρες να εγκρίνουν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ε, πληρούν τα αριθμητικά κριτήρια σύγκλησης πριν ε, περάσουν στο ευρώ. Αυτά τα βήματα όμως δεν αρκούν για να ωφεληθούν από τη συμμετοχή στην ε, Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ακούραστες προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν διαχρονικά ούτως ώστε να κάνουμε αντικυκλικά να πάρουμε αντικυκλικά ε, δημοσιονομικά μέτρα, ε, μέτρα μακρό προφύλαξης και πρόληψης, ε, σωστή διαχείριση του χρέους κλπ. Ε, θα πρέπει να δοθεί ε, προτεραιότητα ούτω ώστε να ε, διατηρηθεί ε, η ε, σύγκληση συνεχιζόμενη. Είναι προς το συμφέρον όλων των κρατών μελών να αποφύγουν ασυνέπειες διαχρονικά. Το front loading είναι σημαντικό για να έχουμε οικονομικά ωφέλη. Η αρχή της νομισματικής ένωσης συνοδεύτηκε από έντονη σύγκληση ε, μακροπρόθεσμων ε, επιτοκίων, αλλά πολλές χώρες δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν ε, την άνθηση που δημιουργήθηκε για να βελτιώσουν τα οικονομικά τους. Πολλές από τις χώρες που ήρθαν αργότερα πήραν μέτρα πιο θετικά. Οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωζώνη τώρα θα πρέπει να είναι επαρκώς έτοιμη. Όχι μόνο για το κοινό νόμισμα αλλά και για την τραπεζική Τραπεζική Ένωση. Ένα ε, ε, μέλλον ε, που θέλει να ενταχθεί δηλαδή θα πρέπει να ζητεί στενή συνεργασία μεταξύ εθνικού τραπεζικού επόπτη και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει δηλαδή να γίνει πλήρης αξιολόγηση. Το ερώτημα αν θα επεκταθεί η Ευρωζώνη ε, ε, είναι και θα παραμείνει πολιτική απόφαση που θα λαμβάνεται από τους πολίτες και τους αιρετούς εκπροσώπους του. Παράλληλα, οι οικονομικές και νομικές προϋποθέσεις και συνθήκες για την επιτυχή συμμετοχή απαιτούν ε, εντελεχή έλεγχο προς το συμφέρον όλων των μερών. Ολοκληρώνω. Αντί να ε, επιχειρηματολογούμε για το αν είναι πιο σημαντικό να διευρυνθεί ή να εμβαθυνθεί η Ένωση. Εγώ λέω σήμερα ότι οποιαδήποτε διεύρυνση της Ευρωζώνης θα πρέπει να εμβαθυνθει η ενωση εγω λεω σημερα οτι οποιαδηποτε διευρυνση τη ευρωζωνη θα πρεπει να συνοδευεται με, από μέτρα εμβαθυνση και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο. Τα κοινοβούλια έχουν ένα κρίσιμο ρόλο να παίξουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια μπορούν να προωθήσουν την νομοθετική ολοκλήρωση. Μπορούν να ε, ε, δουν ούτω ώστε να υπάρχουν ε, να, να, να παρακολουθούν μήπως ε, υπάρξουν ανεπιθύμητες επιρροές εθνικών πολιτικών ε, και, και να παρακολουθούν τους ευρωπαϊκούς δρόντες και τις εθνικές κυβερνήσεις που είναι υπόλογες για τις δράσεις τους στην ΟΝΕ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα έχετε ζητήσει ε, να πάρετε το λόγο και θα ξεκινήσουμε με την κυρία Κρέτσου από τη Ρωμανική Γερουσία. Σας θυμίζω σε όλους πως έχετε δύο λεπτά για την παρέμβασή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμμετείχα σε, στη συνέλευση άρθρου 13 εξ αρχής. Με κίνδυνο να γίνω κουραστική, θα επαναλαμβάνω διαρκώς ότι εξισορρόπηση των ε, λογαριασμών είναι πιο υγιής για την ευρωπαϊκό νόμισμα και την ευρωπαϊκή οικονομία παρά ο ισολογισμός όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά. Οι θεσμικές φωνές ζητούν τώρα ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. η έκθεση η σχετική λέει ότι η εξισορρόπηση των πλεονασμάτων χρειάζεται επιγόντως και θα ήταν ωφέλιμη για όλους. Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχής γιατί είχα δίκιο. Αλλά όμως η πρόταση αφορά μόνο την Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι φροντίζουμε το νόμισμα αλλά δεν φροντίζουμε καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να μείνουν δηλαδή τα, οι χώρε που δεν ανήκουν στο ευρώ τουλάχιστον να είναι μέσα στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Τα κάτι μελη που δεν είναι ακόμα μέλη της Ευρωζώνης είναι μέρη της ενιαίας αγοράς με υψηλά επίπεδα ολοκλήρωσης και ωφελούνται από μια προσωρινή εξαίρεση από το ευρώ σημαντικά ποσοστά των ευρωπαϊκών κεφαλαίων στους τραπεζικούς τους τομείς και έχουν ως βασικούς εμπορικούς εταίρους τους ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Αυτά τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να πέσουν θύματα κρίσης όπως και τα μέλη της Ευρωζώνης χωρίς να μπορούν να ωφεληθούν από τους μηχανισμούς ε, που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού προπολογισμού και από τους κανόνες που έχουν δημιουργηθεί για να βοηθηθούν όσοι έχουν προβλήματα. Αυτό το χάσμα, ο διχασμός ανάμεσα στο εκείνους που είναι στο ευρώ και εκείνους που δεν είναι θεωρείται ως ε, απορριπτικός και ενισχύει τους ευρωσκεπτικιστές. Είναι επικίνδυνος εκτός αν σκεφτούμε ότι μπορεί να σωθεί το ευρώ χωρίς την Ένωση. Εγώ δεν το πιστεύω. Το ευρώ είναι το έμπιστο νόμισμα, ε, αξιόπιστο νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί παγκοσμίω να ισχυροποιηθεί μόνο αν ενεργήσουμε ώστε να διατηρήσουμε ψηλή εμπιστοσύνη στην Ένωση και στο ευρώ. Σας ευχαριστώ και ε, ο κύριος ε, Περμενών από την Λετωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κύριο θέμα της συζήτησης είναι η οικονομική διακυβέρνηση της, Ευρωπα... της Οικονομικής Ένωσης. Στρατηγική αναθεώρηση του ε, Δημοσιονομικού Συμφώνου και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι αυτά η προτεραιότητα για να καθορίσουμε την ε, παραγωγή και την μείωση του διαθετικού ε, λίματος. δεν θα πρέπει να γίνουν λάθη στρατηγική. Θα πρέπει να βρεθούν ε, λύσεις όσον αφορά τις, τον κανόνα περί δαπανών. Οι δαπάνε είναι άμεσα υπό τον έλεγχο των κυβερνήσεων. Έπειτα ο υπολογισμό δυνητική ανάπτυξη και η μείωση του διορθωτικού ελλείμματο θα πρέπει να βασίζονται σε μακρύτερο χρονικό διάστημα από ότι τα δύο έτη που χρησιμοποιούνται τώρα. Τριετία ή τετραετία είναι προτιμότερη. Τρίτον, ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη θα πρέπει να επεκταθεί εξαιρώντα την εθνική συγχρηματοδότηση ε, των προγραμμάτων των, ταμείων, των διευθυντικών ταμείων τη Ένωση, δημοσίων ε, ε, επενδύσεων από τον υπολογισμό του ελλείμματος έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις για την παιδεία, την υγειονομική περίθαλψη, τις ψηφιακές υποδομές και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ο νέο ρόλο τη δημόσια οικονομία θα πρέπει να είναι κατευθυντήρια γραμμή για την δημοσιονομική πολιτική, έτσι ώστε στον οικονομικό κύκλο κάθε κυβέρνηση να μπορεί να διανυστεί μόνο για να επενδύσει και όχι για να χρηματοδοτήσει τι τις τρέχουσες δαπάνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δικαιοσύνη και οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη θα πρέπει να διευκολύνουν και να στηρίξουν τον υψηλό όγκο δημοσίων επενδύσεων που απαιτούνται ώστε να στηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι θέμα κλειδί για την ύπαρξη και το μέλλον της Ένωσης. Εάν η δημοσιονομική πολιτική δεν αλλάξει, πραγματικά θα αποτύχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Now... Σας ευχαριστώ. Και τώρα είναι η σειρά ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αλφρέτ Σάντ. Ευχαριστώ. Είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να συζητήσουμε την πρόοδο της Ευρωζώνης ε, από μια στρατηγική προοπτική γιατί μας αποκαλέσαν τεχνοκράτες ε, και κάθε βήμα που γίνεται μπροστά εξαρτάται από το τι γίνεται αλλού. Φαίνεται όσο, συμβαίνουν εδώ να είναι σε διαφορετικό πλανήτη. Τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια δεν συμμετέχουν σε όσα συμβαίνουν. Η Τραπεζική Ένωση λειτουργεί επί τόπου, ενώ η Ένωση Κεφαλαγοράς υπαναχωρεί και ε, το μεταξύ τα εθνικά ελλείμματα είναι υποέλεγχο. Όμως η ανάπτυξη της Ευρωζώνης δεν ε, είναι θεαματική. Το project της Ευρωζώνης είναι κυρίως πολιτικό, αλλά έχει γίνει ουσιαστικά ένα ε, παιχνίδι σκακιού για τους ε, τεχνοκράτες και ε, μπορεί να υπάρχουν δύο τρόποι να βγούμε από αυτό τον κύκλων ε, ε, να δεκτούμε ότι υπάρχουν νικητές και ιτεμένοι για την Ευρωζώνη, να δούμε πού έγιναν οι ήτες και αν υπάρχουν πολιτικοί τρόποι να τις αντιμετωπίσουμε και να έχουμε πιο ισορροπημένο αποτέλεσμα. Τότε μπορούμε να οικοδομήσουμε και δομές για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία. Αυτές οι προτάσεις που ακούστηκαν κυκλοφορούν εδώ και καιρό. Αυτό θα ε, βοηθούσε την Ευρωζώνη να αναπτυχθεί, όμως όποτε φαίνεται θα γίνει. Το δεύτερο θα είναι να συνεχίσουμε την τεχνοκρατική τάση που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Ε, Όμω, οποιοδήποτε βήμα προ τα μπρο ενδεικνύεται χωρί ε, να ακούτε τι λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, δεν θα γίνουν τελικά περισσότερα, αλλά όταν η επόμενη κρίση καταφτάσει, αυτό το μικρό βήμα προς τα μπρος θα μπορούσε να μας σώσει για να χαράξουμε νέες αρχές. Διαφορετικά είμαστε χαμένοι. Η επόμενη κρίση θα μας βρει μη προετοιμασμένους. Ε, το να τα ε, ανακατεύουμε και να έχουμε διάμεσες λύσεις είναι μια ε, επιλογή των Βρετανών. Όμως τώρα το Brexit έχει ήδη λάβει χώρα. Ευχαριστώ κύριο Στούζεκ από το Κρατικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα μιλήσω κρατικά. Η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγκυται κυρίως σε κανόνες. Στην τελευταία δεκαετία πολλά έγιναν για την απλούστευση και ενίσχυση των κανόνων, κυρίως των δημοσιονομικών κανόνων μέσω του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και μέσω της υλοποίησης του Δημοσιονομικού Συμφώνου ως ε, τμήμα ε, της σταθεροποίησης και της διακυβέρνησης δημοσιονομικής σταθερότητας ε, στο ΙΝΟΝΕ δεν υπάρχει σύστημα δημοσιονομικών μεταφορών για κράτη ή περιοχές που αντιμετωπίζουν ασύμετρα μικροοικονομικά σοκ. Αυτή η αδυναμία φάνηκε κατά την τελευταία κρίση όταν ε, κάποιες από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο βίωσαν σοβαρή ύφαση χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταφορών κονδυλίων από τον κοινό προπολογισμό. Γι' αυτό εγώ χαιρετίζω το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ε, ως ένα μέσο που παρέχει βοήθεια στα κράτη που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Επίση, η διαδικασία αντιμετώπιση μακροοικονομικών ισοβεριών θα μπορούσε να ενδυναμώσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, το μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται για ένα διορθωτικό μηχανισμό για τα κράτη-μέλη που έχουν μεγάλε ανισορροπίε. Τα κράτη που αρνούνται να εφαρμόσουν σημαντικέ συστάσει θα μπορούσαν να τεθούν στο διορθωτικό σκέλο τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο. Ένα άλλο διαβλό ε, για να πετύχουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση είναι η Ένωση Κεφαλαιογορών, τη οποία υλοποίηση εκκρεμεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σλουτίκ από τις κατοχώρες. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση για τον κύριο Σεντένιο. Διάβασα το tweet του όπου απαντούσε σε ένα tweet του Υπουργού μας των Οικονομικών, του κυρίου Χουκστρά, για τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το Ολλανδικό Κοινοβούλιο στη διαφάνεια του Eurogroup. Ο κύριος Σεντένιο έκανε tweet ότι ε, τα ε, ε, ελήφθησαν μέτρα και η διαφάνεια ε, κατοχυρώνεται σταδιακά. Ποια είναι τα νέα βήματα που θα λάβετε το 2020 για τη βελτίωση της διαφάνειας και μπορείτε να μας σχολιάσετε το κείμενο του συναδέλφου Πίτερ Όμσεχτ ε, σχετικά με κάποιες προτάσεις για ταχύτερο άνοιγμα των εγγράφων που ε, καταρτίζει ε, το Συμβούλιο Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Πισλάρου, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι λιγότερο απεσιόδοξη για το μέλλον, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ε, μείνουμε στο σημερινό φόβο. Γι' αυτό κάνουμε το, την πράσινη συμφωνία για τον το ψηφιακό μετασχηματισμό. Το ίδιο θα γίνει και με την ΟΝΕ. Ε, είναι γεγονός ότι υπάρχει νομική υποχρέωση ε, ένταξη στο ευρώ. Δεν είναι κάτι ε, προαιρετικό αυτό. Έχουμε χώρες ε, που θέλουν και είναι έτοιμοι, άλλοι θέλουν αλλά δεν είναι έτοιμες και έχουμε και χώρες που είναι έτοιμες αλλά δεν θέλουν να μπουν στο ευρώ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τις χώρες αυτές προσπαθώντας να κάνουμε περισσότερα για να ενημερωθούν οι πολίτες και αυτό δεν είναι τεχνοκρατικό θέμα, είναι πολιτικό. Για τις χώρες που δεν είναι έτοιμες εκεί θα χρειαστεί βοήθεια και πρέπει να πιέσουμε την ε, διαδικασία μετά τον Brexit, θα πρέπει να συνενωθούμε περισσότερο. Αυτό πρέπει να είναι ένα ε, εγχείρημα για το μέλλον. Ε, Είμαι ε, για το πρόγραμμα ξένων επενδύσεων στη σχετική έκθεση και πρέπει να πω ότι χαίρομαι διότι θα έχουμε κάποια μέσα που θα δημιουργήσουν κίνητρα. Έχουμε την νομική υποχρέωση αλλά τώρα δημιουργούμε και κίνητρα για την ένταξη στο ευρώ. Η διαδικασία λοιπόν διεύρυνση και εμβάθυνση ε, συνοδεύονται από εργαλεία. Αλλά πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία και να έχουμε διαφανή τρόπο να λειτουργεί το μέσο, να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε υπόλοιποι ψυχολόγοι για λογοδοσία στους πολίτες μας. Τέλος, όσο νέος ε, συντονιστής ε, για την έκθεση για την απασχόληση, θα πρέπει να πω ότι η σύγκληση είναι κλειδί. Η πραγματική ε, σύγκληση. Όταν μιλάμε για ψηφιακό μετασυμματισμό, πράσινη συμφωνία, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια κοινωνική επένδυση, κοινωνική συμφωνία. Επενδύσεις στη στέγη, στο ε, ε, ψηφιακό γραμματισμό κλπ. Έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μία βιώσιμη διεύρυνση της ε, Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Σλαλόβατσα από το Κρατικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές και ευρωβουλευτές. Η ε, κρίση έπεισε για την Τραπεζική Ένωση τη δημιουργία νέων μηχανισμών. Ε, θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να περάσουν αρμοδιότητες ε, που αφορούσαν το τραπεζικό τομέα. Η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης όμως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να ολοκληρωθεί με το σύστημα προστασίας των καταθέσεων και ε, μέτρα ασφάλισης κινδύνου. Η Τραπεζική Ένωση ε, πρέπει να ε, ολοκληρωθεί και θα πρέπει να υπάρχει και backstop ούτως ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Εκτός της Τραπεζικής Ένωσης χρειάζεται και η Ένωση Κεφαλαίου Αγορών ο μιλητής παρακαλείται να μιλά αργότερα. Οι διερμηνείς ζητούν συγγνώμη γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εύκολα την ταχύτητα του ομιλητή. Το νομοθετικό πλαίσιο για την σύσταση της Επιτροπής της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών είναι πολύ ευρύ. Ε, προβλέπει ε, πλαίσιο για πτωχεύσεις, διασυνοριακές επενδύσεις. Εμείς χαιρόμεθα ε, για τις συστάσεις του Συμβουλίου και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι οι συστάσεις για την Ευρωζώνη καλούν την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών και προωθούν όλα τα θέματα οποία θα διευρύνουν και θα εμβαθύνουν την ΟΝΕ. Ο κύριος Κόσορ από το Κροατικό Κοινοβούλιο πιστεύω. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πέρα από τις ε, θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να ενδυναμώσουμε και την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γι' αυτό τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων και των νέων μηχανισμών. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε μηχανισμούς συντονισμού και να έχουν κυριότητα των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω εμβάνθυνση της ΟΝΕ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και την Τραπεζική Ένωση, να συστήσουμε την Ένωση Κεφαλαγορών και να έχουμε και μηχανισμούς προστασίας σε επίπεδο βρεζόνης. Σε ό,τι αφορά την πρόοδο της Κροατίας. Έχουμε μειώσει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και στείλαμε μία επιστολή προθέσεων για να ενταχθούμε στο μηχανισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό ε, μας βοήθησε επειδή είχαμε συζητήσεις ε, με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν και το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων τα θεσμικά όργανα έδειξαν την πολιτική τους βούληση να διευρύνουν την Ευρωζώνη. Στην επιστολή η Κροατία ε, θα υιοθετήσει 90 μέτρα σε έξι τομείς, θα ενδυναμώσει την συνεργασία με την ΕΚΤ, θα ενισχύσει το μακρό προληπτικό πλαίσιο, θα καταπολεμήσει την νομοποίηση παράνομων εσόδων, και θα βελτιώσει τη συλλογή και ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων, θα βελτιώσει τη διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα και θα μειώσει το διοικητικό άχθος. Η Κροατία θέλει να πετύχει τους στόχους αυτούς μέχρι τα μέσα του 2020 και αυτό θα δείξει ότι είναι σοβαρός υποψήφιος για να ενταχθεί στον ERM. Σε ό,τι αφορά την οικονομική διακυβέρνηση, θα πρέπει να φέρουμε πολιτική ευθύνη και στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικός ο ρόλος των κοινοβουλίων. Ευχαριστώ. Thank you very Now, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαυρίδης από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Έχω την άποψη ότι η πραγματική σύγκληση των οικονομιών μας είναι η καλύτερη υπηρεσία προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα και ταυτοχρόνως είναι η καλύτερη απάντηση που έχουμε στους λαϊκιστές και σε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό όραμα. Αν το συμμεριζόμαστε αυτό, δηλαδή ότι θα πρέπει να έχουμε πραγματική σύγκληση των οικονομιών μας, θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα και να βρούμε εκείνα τα εργαλεία τα οποία στην πράξη θα μας φέρουν κοντά γιατί εμένα είναι η δεύτερη μου θητεία και ομολογώ ότι ορισμένες φορές έχω ακούσει τα ίδια πράγματα τόσες φορές που αισθάνομαι ότι έχω κουραστεί. θα πω ένα δυο παραδείγματα. σε σχέση με το ευρωπαϊκό εξάμεινο κάτι συγκεκριμένο προτείνουμε ως πολιτική ομάδα εδώ και χρόνια κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια να συμπεριληφθούν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο δεύτερον σε σχέση με τη δομή και την εμβάθυνση κάποιων από τα οικονομικά εργαλεία στην οικονομική νομισματική ένωση δεν μπορώ να φανταστώ ως οικονομολόγος ότι μιλάμε για εμβάνθηση της κοινή ευρωπαϊκής αγοράς και ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση. πώς είναι δυνατόν κατανοώ τα τεχνικά προβλήματα αλλά να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα το κύριο εμπόδιο ήταν και παραμένει η πολιτική εναντίωση συγκεκριμένων κρατών. δεύτερο και το τελευταίο μου σημείο είναι το εξή σε σχέση με την μετάβαση στον στόχο του 2050 τονίζω δύο λέξεις δίκαιη μετάβαση και ρεαλιστική προσέγγιση. αυτό είναι θεωρώ η καλύτερη οδός σε όσους συμμεριζόμαστε το ευρωπαϊκό εγχείρημα γιατί οποιαδήποτε ταρακούνησή του μπορεί να μας δημιουργήσει και νέα προβλήματα στην πορεία μας για το κοινό μας όραμα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τώρα ο κύριος από το Bundestag. Αξιότιμοι πρόεδροι, η δομή είναι διακυβερνητική βάσει διεθνών συμφωνιών. Η σημερινή συζήτηση ε, γίνεται ε, για το πέρασμα στο ενωσιακό δίκαιο από τις κρατικές συμφωνίες. Πρέπει οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων να είναι δημοκρατικές, χρειάζεται προσοχή και πρέπει να έχουμε υπόψη και τη σημασία των εθνικών κοινοβουλίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για προϋπολογισμό και θέματα φορολογίας. Η αναθεώρηση του 2 και 6 ε, είναι σημαντική. Η, ε, μετά την κρίση θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ούτως ώστε να έχουμε ε, συντονισμένες διαδικασίες για χώρες που ε, ε, υπέφεραν από την κρίση ή αντιμετωπίζουν κρίση. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε το θέμα των επενδύσεων. Η πρώτη μεταρρύθμιση θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό ισχύει και για το Common Backstop, αλλά οι κίνδυνη των ε, ισολογισμών των τραπεζών θα πρέπει να είναι πάντοτε ε, στο στόχαστρό μας. Πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις το BIC είναι πολύ σημαντικό βήμα προς το μέλλον και η ανταγωνιστικότητα των ε, οικονομιών μας θα πρέπει να ε, παρουσιάσει σύγκληση σημαντικό είναι να αποφευθούν επικαλύψεις ε, επίσης το υπενθυμίζω τα 280 δις ευρώ υπόλοιπο προς διάθεση προς εκαθάριση ε, είναι σημαντικό επίσης να ε, ε, έχουμε επαρκή διακυβερνητικά μέτρα στα πλαίσια της διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βότσης από την Κύπρο. Ομολογουμένω, η τρέχουσα δημοσιονομική αρχιτεκτονική σχεδιάστηκε ω απάντηση στην πρωτοφανή οικονομική κρίση του 2008 και συνεπώ χρήζει αναπροσαρμογή προκειμένου να ανταποκρίνεται στι σύγχρονε προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ένωση και στου φιλόδοξου στόχου που έχει θέσει για οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η απλοποίηση τη τρέχουσα δημοσιονομική δομή, η ενίσχυση τη διαφάνεια της εμπιστοσύνης των πολιτών της πολιτικής υπευθυνότητας της αξιοπιστίας των δημοσιονομικών κανόνων είναι κρίσιμη σημασία για περαιτέρω διεύρυνση και βάθηση τη δημοσιονομική διακυβέρνηση τη Ευρωζώνη. Το πιο σημαντικό όμω, και με αυτό θα τελειώσω την παρέμβασή μου, είναι η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασφάλιση Καταθέσεων, που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση τη Τραπεζική Ένωση και την αποκατάσταση της θεμελιώδους αρχής της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης. Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων είναι καταλητική σημασίας για τη διασφάλιση της ισότιμης προστασίας των καταθετών ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης και για άρση του σημερινού παράδοξου όπου η δημοσιονομική εποπτεία και εξυγίαση επιτελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ η προστασία των καταθετών παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να καυστηριάσω το γεγονός ότι οι κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχία και εξυγίασης και τα επώδυνα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο των προγραμμάτων, των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, η χώρα μου η Κύπρος τα έχει ζήσει καλά στο πετσί και ο Κυπριακό λαός, υλοποιήθηκαν με τη μορφή του κατεπήγοντος ενώ η πρόοδο όσον αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού συστήματο ασφάλισης καταθέσεων είναι εξαιρετικά αργή δεδομένου ότι η υλοποίησή τη εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί αν θα επιτευχθεί μετά το 2024. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Now, uh, Ευχαριστώ. Uh, Κυρία Μάρκες, ο Μάρκες, συγχωρείτε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Στο πλαίσιο αυτής ε, της συζήτησης οικονομικής διακυβέρνησης θα ήθελα να αναφέρω αρχικά ότι αν η νομισματική πολιτική θα πρέπει να σώσει το ευρώ σε ευλογό χρόνο είναι γιατί οι κανόνες ε, και ε, όσα έχουμε σήμερα αναποδείχθηκαν ανεπαρκή και αναποδείχθηκαν ανεπαρκή ακόμη και μετά την ανακοίνωση του 2015 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήθελε να προσδώσει μεγαλύτερη ευελιξία στην ερμηνεία των κανόνων αυτών. Ως, ε, όπως είπε και εδώ ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ, η οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να υποστηρίζει την ανάπτυξη και εγώ θα έλεγα την βιώσιμη ανάπτυξη ταυτόχρονα να συνεισφέρει έτσι ώστε να έχουμε υγιή δημόσια οικονομικά. Η οικονομική, οικονομική ανάπτυξη γίνεται κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λόγω ε, του ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην καινοτομία δεν επαρκεί αλλά επίσης υπάρχει και μία τάση ε, σε, στο ότι επικεντρώνονται σε μια λογική εξοικονόμησης. Οι κυβερνήσεις χρειαζόμαστε κανόνες που να υποστηρίζουν τις επενδύσεις και ιδίως τις πράσινες επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ένα χρυσό κανόνα για την υποστήριξη των πράσινων επενδύσεων. Επίσης χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο πιο ολοκληρωμένο το οποίο θα ε, θέτει μεταξύ των στόχων, μεταξύ των μηχανισμών συντονισμού του στόχους βιώσιμη ανάπτυξη χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία στην οικονομική διακυβέρνηση. Κυρίω να έχουμε κανόνε αντικυκλικού και όχι προκυκλικού όπω είχαμε στο παρελθόν. Θα πρέπει να προχωρήσει ε, ο μηχανισμός σταθεροποίησης με πραγματικό προπαλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πραγματική ένωση τραπεζών ε, και με πραγματικό ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Και θα ήθελα να αναφερθώ και τέλος ε, σε ένα μηχανισμό που αφορά το macroeconomic imbalances procedure. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία αυτή και στις χώρες που έχουν έλλειμμα αλλά και στις χώρες που έχουν πλεόνασμα θέλουμε τελικά να έχουμε μια οικονομία που να μπορεί να εξάγει κάποια στιγμή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταύρου από την Κύπρο. I will speak in my mother tongue. Το τρέχον δημοσιονομικό πλαίσιο συνέβαλε στο στενότερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της Ευρωζώνης, την ενίσχυση της οικονομικής της ανθεκτικότητας σε ενδεχόμενους οικονομικούς κλειδονισμούς και την αναδική σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών, αν και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες προσκλήσεις του κάθε κράτους μέλους χωριστά, το δημοσιονομικό πλαίσιο κατέστη πολύπλοκο, αδιαφανές και αναποτελεσματικό και γι' αυτό χρήζει περαιτέρω εξορθολογισμού, απλοποίησης και αναπροσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα. Δράτω με της ευκαιρίας να χαιρετήσω την πρόσφατη εξαγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διεξαγωγή Δημόσιας δημόσιας διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για το μέλλον του πλαισίου οικονομικής εποπτείας. Φιλοδοξούμε ότι η διαβούλευση θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα συμβάλλοντας την κριτική αξιολόγηση, την αποτίμηση και την αναβάθμιση του υφιστάμενου οικονομικού πλαισίου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στους φιλόδοξους της για ψηφιακό και οικολογικό μετασχηματισμό καταλήγοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω τον καταλυτικό ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν τα εθνικά κοινοβούλια μέσω της ενίσχυσης του εποπτικού τους ρόλου στη διαδικασία του ευρωπαϊκού εξαμήνου στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας και στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας του πλαισίου δημοσιονομικής διακυβέρνησης. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουίτζι Ματρατίν από την Ιταλία. you. Ε, για το BIC. Έτσι όπως διαμορφώνεται, μου φαίνεται ότι μοιάζει σαν ε, ε, διαρθρωτικό ταμείο που θα στηρίζεται από τα κράτη. Αυτό που χρειαζόμαστε, αυτό που χρειάζεται και αυτό που λείπει από την ολοκλήρωση είναι η σταθεροποίηση, η, μια λειτουργία σταθεροποίησης η οποία θα επιτυγχάνεται από ένα πρόγραμμα προστασίας της απασχόλησης για να καλύψει και τα προβλήματα εφαρμογής που έχουν να κάνουν και με ε, ε, δαπάνες αν θέλουμε σταθεροποιητικό αποτέλεσμα στον ενωσιακό προϋπολογισμό θα πρέπει να δούμε τις ελλείψεις εφαρμογής που έχουν να κάνουν με την έλλειψη επενδύσεων. Ο καλύτερος τρόπος ε, κάλυψης και προστασίας από ασύμετρα σοκ. Ε, Επίση, η δημοσιονομική ικανότητα είναι σημαντική. Επίσης, γιατί δεν επεξεργαζόμεθα αποτελεσματική ανταλλαγή μεταξύ ε, κάποιων ορίων σε σχέση ε, με το χρέος και τα στοιχεία του ενεργητικού ε, με βάση το χρέος, το, το κρατικό, το δημόσιο χρέος ε, να επεξεργαστούμε έτσι κάποια αποτελεσματικά όρια ε, ούτως ώστε να ε, βελτιώσουμε και τους ισολογισμούς των εμπορικών τραπεζών και επίσης ας, έτσι θα λύσουμε και το πρόβλημα που έχουμε με τις εκροές. Ας δούμε ε, που είναι η πηγή των εξωτερικών στοιχείων, το επίπεδο και η δυναμική του δημόσιου χρέους. Ε, ε, το εξωτερικό στοιχείο, αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος των δημοσιονομικών κανόνων. Θα σταματήσουμε τώρα να παίρνουμε ερωτήσεις, γιατί αλλιώς δεν θα τις προλάβουμε όλες. Δίνω το λόγο στον κύριο Ταντέσκι από την Πολωνία. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Επίτροποι, συνάδελφοι, η Πολωνία είναι υπέρ του προγράμματος στήριξης των μεταρρυθμίσεων, όπως στηρίζουμε άλλωστε και το δημοσιονομικό μέσον για την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα. Θέλουμε περισσότερε μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα από χώρε εκτό Ευρωζώνης. Είναι πολύ σημαντικό για να προωθήσουμε την οικονομική του σύγκληση με τις χώρες Ευρωζώνης. Η Πολωνία είναι υπέρ των κάτωθη. Όταν πρόκειται για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και του προπολογισμού για αυτά τα μέσα, πρέπει να τηρήσουμε τα ποσά που προτάθηκαν το Δεκέμβριο του 2019. 2 3 αυτό το, ε, την αναλογία. Θέλουμε επίσης συνοχή μεταξύ των μέσων για την Ευρωζώνη και των μέσων για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Πιστεύουμε ότι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον αντίκτυπο ε, των ε, επιμέρους κρατών και το πακέτο μεταρρυθμίσεων που προτείνει η Επιτροπή για να υπάρχει κάποια δημοσιονομική αυτονομία. Η Πολωνία χαιρετίζει το γεγονός ότι οι προτινόμενες λύσεις προκειμένου περί αυτών των προγραμμάτων ευθυγραμμίζονται με την, τις αρχές της οικονομικής διακυβέρνησης ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Πολωνία πιστεύει ότι οι εσδήποτε νέες δράσεις θα πρέπει να στηρίζουν τη σύγκληση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επιμέρους κράτη-μέλη. Δεν πρέπει να εμβαθύνουμε τις ε, διαιρέσεις που υπάρχουν σήμερα εντός της, Ευρωζω... της Ένωσης. Ευχαριστώ. Mr. Di Fazio, which is the rapporteur for the European Economic and Social. θα δώσουμε το Πιστεύω πως ε, είναι σημαντικό να βασιζόμαστε στην ε, σταθερότητα και την ε, ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο όμως είναι σημαντικό να βασίζεται σε μία μακρόπνοη στρατηγική. Αυτό νομίζω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μία μακρόπνοη στρατηγική θα πρέπει να προβλέπει τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το Πράσινο Σύμφωνο ε, και τον αντίκτυπο αυτού στον κόσμο της εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο. Θα είναι σημαντικές λοιπόν τα βοηθήματα που θα δοθούν και ο συντονισμός της διακυβέρνησης μέσω των δημοσίων επενδύσεων όσον αφορά τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και στην ε, εκπαίδευση που θα μπορέσουν να δυναμώσουν και μέσω της βοήθειας προς τη τις ε, δημόσιες ιδιωτικές επενδύσεις και τα κίνητρα όπως ήδη έχουμε στην Ευρώπη, ιδιωτικές επενδύσεις μέσω ε, δημοσίων ε, εγγύσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά σημαντικό και το έχουμε ήδη πει ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης να αναθεωρηθεί και ήδη το καλεί αυτό η Κομισιόν αναθεώρηση της διακυβέρνησης. Εμείς ε, θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η αναθεώρηση και άκουσα με μεγάλη προσοχή τα όσα είπε ο Επίτροπος Τζεντιλόνη ότι δεν θέλουμε να έχουμε πιο ε, ε, ισχυρούς κανόνες ή περισσότερους κανόνες. Θέλουμε να τους εξυγχρονίσουμε όμως έτσι ώστε να έχουν ε, αποτέλεσμα και επιρροή στο μέλλον μας. Και γι' αυτό θα είναι σημαντικό να εξετάσουμε και τους κοινωνικούς πυλώνες αλλά και να έχουμε και μια ιδιαίτερη βοήθεια από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών τόσο εδώ στις Βρυξέλλες μέσω της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της συμβουλευτική της, ε, λειτουργία, όπως και στις χώρες όπου θα πρέπει να βοηθηθούν για την υλοποίηση της διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα προχωρούμε στην κυρία Μάρκες του Ευρωκοινοβουλίου. Εγώ θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα να πω το εξή, να ευχαριστήσω για όλες τις ε, ομιλίες από τους προσκεκλημένους μας. Αυτή η συζήτηση ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε τέτοιες ε, διακοινοβουλευτικές ε, διασκέψεις από την πλευρά των Εθνικών Κοινοβουλίων και όντω οι συζητήσεις αυτές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε και να μοιραστούμε από υπόψη, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε διαφορετικέ αρμοδιότητε, αλλά ε, και, δύο κοινοβούλια, δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, συμβάλλουμε για τον καθορισμό των ευρωπαϊκών πολιτικών. Ήθελα να κάνω τρει σύντομε παρατηρήσει. Η πρώτη, σε σχέση με την ευάθυνση τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης το 2017 στη Ρώμη, με την επέτειο τη συνθήκη τη Ρώμη, ο Πορτογάλος Πρωθυπουργό είπε ότι δεν θα έχει νόημα η της Ρώμης αν δεν αφαιρόταν στην ευάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, έχουμε παρακολουθήσει την εξέλιξη των πολιτικών αποφάσεων σε αυτό το τομέα και οι πολιτικές αποφάσεις ήταν πολύ αργές. Ερώτησή μου λοιπόν είναι, ποιο, ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά με το τελευταίο οδικό χάρτη που υιοθετήθηκε σε σχέση με τη συμπεριφορά της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Τώρα, δεύτερη παρατήρηση όσον αφορά το Πράσινο Σύμφωνο Στατηγική Οικονομικής Ανάπτυξης. Για να εισάγουμε το Πράσινο Σύμφωνο στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας, ε, χρειαζόμαστε δύο βασικά θέματα στη μεταβατική περίοδο. Το πρώτο είναι περισσότερη ευελιξία και όπως γνωρίζουμε περισσότερη ευελιξία σημαίνει περισσότερη περιπλοκότητα αλλά Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε ένα σύμφωνο πιο απλό. Οπότε θέλω να ρωτήσω πώς θα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, αυτούς τους δύο στόχους, ευελιξία και απλότητα. Τέλος, ως εισηγήτρια για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο του Eurogroup που ξέρω πως ήδη αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα στην αρχική του ομιλία τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το δημοσιονομικό μέσο για τη σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα μέσα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για, μέχρι το 2027. Ευχαριστώ πολύ και ως πέσκο από την Ιταλία. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και πρώτα εσάς πρόεδρε την άλλη για όλες σας τις Θέλω να τον τονίσω τα, τα νέα στοιχεία που αναφέρθηκαν εδώ, ε, δηλαδή του ίδιου πόρου για να χρηματοδοτηθούν οι μεταρρυθμίσει. Πρέπει να πω το εξή. Προσοχή, γιατί ήδη οι πόροι μπορεί να ε, ε, προσκρούσουν στι φορολογικέ αρμοδιότητε των χωρών. σω θα πρέπει λοιπόν να βρούμε διαφορετικού τρόπου χρηματοδότηση, όπω α πούμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή τα ευρωομόλογα, όπω α πούμε για το περιβάλλον. Γιατί να μην σκεφτούμε ευρωομόλογα που στόχο θα έχουν την προστασία του περιβάλλοντος, ε, παραδείγματος χάρη. Ε, ο κύριος Σεντένο τον έφερε αυτό και γι' αυτό απευθύνω σε εκείνο την ερώτηση. Μιλήσατε για την ε, νομισματική πολιτική και βεβαίως ελέγχθηκε ο πληθωρισμός, έχει μείνει πολύ χαμηλός, αλλά δεν έχουν γίνει πολλά όσον αφορά την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη. Ίσως αυτό να οφείλεται στις δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες ίσως να μην ήταν στο ύψος των περιστάσεων και τώρα θέλω να στραφώ στον κύριο Πανέτα. Ίσως γι' αυτό τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να αυξηθεί η νομισματική βάση ίσως να μην έφτασαν και στην πραγματική οικονομία. Στην Ιταλία η οικονομία μας βασίζεται στις μικροεταιρείε. Μικροεπιχειρήσεις δεν είναι εύκολο να περάσουμε από τι μικροεπιτερίε στις μεγάλες, ομίλου. και ε, αυτή η προσπάθεια λοιπόν δεν έφτασε στις μικρές εταιρείε. Ίσως θα πρέπει να βρούμε χρήσιμες ε, τρόπους για να βοηθήσουμε την πραγματική οικονομία. Ίσως κάτι πολύ φιλόδοξο να είναι, αλλά ίσως θα έπρεπε να ξαναδούμε και την ε, αποστολή, την εντολή της ΕΚΤ που στόχο έχει να κρατά χαμηλά τον πληθωρισμό, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και την απασχόληση. Τώρα, ευχαριστώ τον κύριο Ντομπρόφσκης που μίλησε για την ε, οδηγία την Μπέιρντε που βασίζεται στο Μπέιλιν, δηλαδή στη χρήση των ε, χρημάτων των αποταμιευτών για να σωθούν οι τράπεζε. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Όσο περισσότερο δεσμευτικοί είναι οι τραπεζικοί κανόνε, τόσο μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα για του πολίτε. Δηλαδή, δεν φτάνουν οι πόροι στην πραγματική οικονομία και γι' αυτό υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, το ε, Μιλήσαμε για Τραπεζική Ένωση και για Ένωση αγορών. Στην Ιταλία διαρκώ αναφέρονται αυτά, όμω πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πω υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Κυρίω στην Ιταλία έχουμε το Ταμείο για τη Διάσωση των ε, Νοικοκυριών. Ε, κύριε Πέσκο, παρακαλώ τη σύντομα. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Γκαραμπάλια από την Ιταλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ταχύτατε ερωτήσει. Ε, ο υπουργό Κουαλντιέρη και ο Πρωθυπουργό μα πριν κάποιες εβδομάδες ε, είπαν για ε, την δυνατότητα να έχουμε επενδύσεις. Όμως από ό,τι καταλαβαίνω έχει κλείσει το θέμα. Δεύτερον, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα και στην Ιταλία και σε όλη την Ευρώπη για ανεμική ανάπτυξη. Φέτος θα είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα και πριν από την κινέζικη κρίση το τελευταίο τρίμηνο έκλεισε πολύ άσχημα και φέτος ε, θα έχουμε μηδενική ανάπτυξη αν πάνε καλά τα πράγματα. Το πραγματικό πρόβλημα αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπόθηκε πριν ότι θέλετε να κάνετε κάτι για να βοηθήσετε. Όμως ε, σήμερα ούτε ένα σέντς δεν φτάνει εδώ στην πραγματική οικονομία και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε γι' αυτό. Μάλιστα, ο κύριος Μικελέφ από τη Μάλτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς ε, μπορούμε να σταθεροποιήσουμε το νόμιμεσμά μας, αλλά δεν θα σώσουμε τίποτα. Δεν θα αντιμετωπίσουμε τις, ε, τα προβλήματα τα κοινωνικά και τα υπερβολοντικά. Σε εθνικό επίπεδο η Μάλτα βλέπει μεγάλη ανάπτυξη στο ΕΠ, αλλά πήραμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αποθεματικά, για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πιθανή κρίση ξεσπάσει. Βεβαίως, όταν λάβουμε υπόψη τις ευρωπαϊκές αρχές αν αλληλεγγύη γίνεται μόνο με νοσηματικούς όρους τότε αυτό δεν είναι ειλικρινές ως το μικρότερο κράτος εγώ περιμένω ένα μέλλον το οποίο θα βελτιώσει την ποιότητα ζωή μας όχι μόνο τα οικονομικά μας Επομένω, ενυπομονώ για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και θα ήθελα επίσης να δω να υπάρχει και μια κοινωνική συμφωνία και χάρη στην κυρία Ντάλη που θα μας βοηθήσει να ενδυναμώσουμε την Ευρώπη αλλά να αλλάξουμε και τον τρόπο που δημιουργούμε τις πολιτικές μας και προβαίνουμε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν θα πρέπει να ξοδέψουμε χρόνο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμούς που θα θέτουν τον Ευρωπαίο πολίτη στο επίκεντρο της καλής διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ένα μεγεθό που ταιριάζει σε όλους, αλλά θα έχουμε ευέλικτου μηχανισμού δημοσιονομικούς που θα επιτρέπει στις χώρες να αναπτυχθούν σε μια ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βαμαμάκη από την Φιλανδία. Στον κύριο Βαμαμάκη, συγγνώμη. Ε, ευχαριστώ. Αλήθεια είναι ότι το σύστημα διακυβέρνησης ε, πρέπει να μεταρρυθμιστεί, αλλά θα πρέπει να μετρήσουμε τους σωστούς παράγοντες, συντελεστές, να το κάνουμε με τρόπο έξυπνο, δηλαδή ανάπτυξη στον τομέα της παραγωγικότητας ε, και Εις ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες, αυτοί βέβαια θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρη. Αν ε, θέλουμε να σώσουμε την ΟΝΕ, τότε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να ισοσκελίζουν τους προϋπολογισμούς, να μειώνουν τα χρέη και να αυξάνουν το, τον ανταγωνι, την ανταγωνιστικότητα. Η εναλλακτική ποια είναι η ε, σύνδεση μεταξύ τραπεζών και χωρών θα ε, διαφοροποιείται. Είναι δύσκολο να υπάρχει συλλογική ευθύνη γιατί οι εθνικές αποφάσεις ε, ίσως αποδυναμώνονται για τις μεταρρυθμίσεις, η Κομισιόν θα έχει μεγαλύτερη εξουσία, αλλά έτσι ίσως επιτευχθούν και στόχοι που με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Πάντως πιστεύω ότι τα, οι, φορείς, ε, οι εθνικοί φορείς λήψεως αποφάσεων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με περισσότερη εμπιστοσύνη. Η κυρία Γιαννάκου ε, από την Ελλάδα. Κυρία Πρόεδρε, ε, το ενδιαφέρον της ε, σημερινής συνάντησης ε, είναι προφανές. Δεν είναι δυνατόν κατά τη γνώμη μου να υπάρξει πραγματικά εμβάθυνση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση χωρίς πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τη γνώμη των κυρίων Σεντένο και Ντομπρόφσκι για το θέμα αυτό λαμβάνοντας υπόψη ότι ανοίγει ένας διάλογος στον ευρωπαϊκό χώρο για την πιθανή τροποποίηση της συνθήκης. Η τροποποίηση της συνθήκης φυσικά δεν θα μπορεί να γίνει αποσπασματικά, να βρούμε τρόπους να παρακάμψουμε αν θέλετε και τις επιθυμίες των πολιτών ή και αν ακούσουμε τις επιθυμίες των πολιτών αυτός να είναι ένας διάλογος χωρίς πραγματικό αποτέλεσμα νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι καταρχήν τα πολιτικά δεδομένα. Τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε. Θέλουμε απλώς να συντηρήσουμε μια κατάσταση με την οποία δημιουργήθηκαν προβλήματα ή μια κατάσταση που δεν ικανοποιεί πλέον ούτε τους πολιτικούς ούτε τους πολίτες ή θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Τότε μας χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική διακυβέρνηση. Μόνο έτσι θα μπορεί να υπάρξει και αντανάκλαση στον οικονομικό τομέα. Είτε αυτό είναι εποπτεία των τραπεζών, είτε είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα οι προσκεκλημένοι μας θα λάβουν το λόγο για σύντομες ε, παρατηρήσεις. Θα ακολουθήσουμε την ίδια σειρά. Δύο λεπτά ο κύριος Δράβκο Μάριτς. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος γιατί είναι πολύ δύσκολο μετά από τόσο γόνιμο και επικοδομητικό διάλογο, συζήτηση, σχόλια που ακούσαμε και ερωτήσεις να απαντήσουμε τόσο σύντομα. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε, θα έλεγα, ότι ε, λάβαμε διδάγματα από το παρελθόν όταν άλλαξα η διακυβέρνηση και έπρεπε να τροποποιηθεί για να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη παγκόσμια ε, ε, χρηματοοικονομική κρίση από τις χώρες μας ο καθένας έχει τις εμπειρίες του, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση είδαμε την ανάγκη επανεξέτασης των δημοσιονομικών κανόνων και της οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σήμερα το πρωί είχαμε στη συνάντηση του ΕΚΟΦΗΝ μια έναρξη αυτής της συζήτησης όπου η Κομισιόν παρουσίασε την πρώτη άποψη έγινε γόνιμος διάλογος και έτσι θα συνεχίσουμε γιατί είναι σαφές από πολλές πλευρές και από τα κοινοβούλια και τα εθνικά και το ευρωπαϊκό ότι δεν υπάρχει μία και μόνο προσέγγιση προς την επίλυση των θεμάτων μας. Όλοι πρέπει να σκεφτούμε τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών δικτών και προφανώς να μην παραμελήσουμε το γεγονός αφού έχουμε κάνει την εμπειρία ότι καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν άρδι, άρδιν προς το χειρότερο. Ε, ευχαριστώ για το διάλογο. Περιμένουμε να συνεχιστεί η συζήτηση για το θέμα αυτό και είμαι βέβαιος ότι σύν το χρόνο θα βρούμε μια ικανοποιητική λύση και ε, αποτελεσματικά μέτρα πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάριος Σεντένο. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Και τις ε, απόψεις σας για την οικοδόμηση της Ευρώπης που όλους μας απασχολεί. Θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις ε, και τέλος θα κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο για το θέμα της ε, συνεδρίασης αυτής. Κύριε Σλότβεκ, αλήθεια είναι ότι η διαφάνεια είναι τεράστια σημασίας για το έργο των δημοκρατικών θεσμικών οργάνων στην Ευρώπη. Είναι ε, εξίσου σημαντικό όπως η ολοκλήρωση. Ε, είχαμε αυξανόμενη διαφάνεια στο Eurogroup, γι' αυτό πρότεινα και έγινε δεκτή η πρόταση να έχουμε ε, κατάθεση εγγράφων που συζητούνται στο Eurogroup, περισσότερη ενημέρωση για το προπαρασκευαστικό σώμα που είναι το Working Group του Eurogroup που είναι τώρα στο website. Επίσης θέλουμε να δημοσιεύουμε τις ημερήσιες διατάξεις και πιο λεπτομερείς συμπεράσματα από τις συζητήσεις. Αυτά τώρα ετοιμάζονται και δημοσιεύονται. Όλα είναι στην ιστοσελίδα τους. Ε, πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι θα συνεχίσουμε να ε, επανεξετάζουμε αυτή την πολιτική στο μέλλον και θα είμαστε έτοιμοι να την βελτιώνουμε. Η πολιτική διαφάνειας τώρα ευθυγραμμίζεται ουσιαστικά με το ΕΚΟΦΗΝ και άλλα συμβούλια και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ε, έχουμε την περαιτέρω ε, ολοκλήρωση, τη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ. Οι οικιέτες ε, θα πρέπει να αποφασίσουν για το νέο μέσο αυτό το BIC, που δεν θα χρηματοδοτείται σε βάρος άλλων πολιτικών. Εγώ εμπιστεύομαι στην ικανότητα των ηγετών μας να εξοπλίσουν αυτό το όργανο με τα απαραίτητα κονδύλια τους απαραίτητους πόρους, ούτως ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του που είναι η σύγκληση και η ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάλτης Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ίσως να επανέλθω σε κάποιες ερωτήσεις που τέθηκαν Καταρχήν για την ε, αναθεώρηση του six pack και του two pack των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ποια είναι τα πιθανά μελλοντικά βήματα. Ένας τομέας που εξετάζουμε είναι η απλούστευση. Και πράγματι ακολουθώντας ε, τις συμβουλές του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου εξετάζουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε από τα κενά και τις διαθετικές ανισορροπίες καθώς ε, ε, είχαμε κάποιους δείκτες ασταθείς και να έχουμε κάποια benchmark τα οποία θα είναι πιο σταθερά. Εργαζόμαστε λοιπόν επί αυτής της απλούστευσης. Επίσης, εξετάζουμε πώς οι μοδιοσημενικοί κανόνες ε, μπορούν να υποστηρίξουν τις επενδύσεις και σε ένα πλαίσιο πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της οικονομίας. Επίσης, είναι σημαντικό να βρούμε τη σωστή ισορροπία, γιατί έχει σημασία και η εφορία. Και θέλουμε και να υπάρχει και συνένεση σε αυτό το τομέα. Έτσι λοιπόν όταν θα συζητάμε για τα επόμενα πιθανά βήματα να έχουμε ένα βαθμό βεβαιότητας ε, ότι θα καταλήξουμε σε μια καλύτερη θέση σε σχέση με σήμερα. Τώρα έχουμε ξεκινήσει μια ευρεία δημόσια διαβούλευση. Ήδη είχαμε μια συζήτηση στο Eurogroup και σήμερα στο ECOFIN. Σήμερα επίσης κάνουμε και τη συζήτηση εδώ. Όμω, όλα τα ενδιαφέροντα μέρη και τα κοινοβούλια είναι πρόσδεκτα να μας δώσουν feedback στη δημόσια διαβούλευση που θα ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του έτους. Πολλά ερωτήματα τέθηκαν σε σχέση με την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Ναι, συμφωνώ ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και να υλοποιηθεί η Ένωση Κεφαλαιογοράων ε, και να έχουμε και δημοσιονομικά μέσα για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση. Από την πλευρά της Κομισιόν εμείς είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε το έργο αυτό τέθηκαν και ερωτήσεις ε, για τη διακυβερνητική φύση κάποιων ε, διευθετήσεων της Ευρωζώνης. Ε, ως Κομισιόν εμείς υποστηρίζουμε το να κινηθούμε προς την κοινοτική μέθοδο Παραδείγματο χάρη, αυτό επιβεβαιώνει την πρότασή μα ε, για να έχουμε την ουσία του Δημοσιονομικού Συμφώνου και στο νομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ο μηχανισμό σταθερότητα να ενταχθεί στο νομοθετικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα τα κράτη-μέλη έχουν επιλέξει να εργάζονται σε μια διακυβερνητική δομή, κυρίω σε ό,τι αφορά και τη μεταρρυθμίση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Όμω νομίζουμε ότι στο μέλλον θα πρέπει να κινηθούμε προ την κοινοτική προσέγγιση. Επίσης, ε, τέθηκαν ερωτήσεις για την πιθανή διεύρυνση της Ευρωζώνης, ε, κυρίως ό,τι αφορά την Κροατία. Συνεργαζόμαστε στενά με τις κροατικές αρχές ε, σε ό,τι αφορά τις πρώτερες δεσμεύσεις για να έχουμε επιτυχή ένδειξη στον ERM2, στο Μηχανισμό Συνολικματικών Ισοτιμιών 2. Επίσης συνεργαζόμαστε με τις βουλγαρικές αρχές ε, σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεργασία με την Κροατία. Θα έλεγα σε σχέση με τις δεσμεύσεις που παρακολουθεί η Κομισιόν είναι γενικά σε καλό δρόμο η Κροατία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Φυσικά υπάρχει και το θέμα της αναθεώρησης του τραπεζικού συστήματος και ίσως η ΕΚΤ είναι καλύτερα να απαντήσει στα θέματα αυτά. Αλλά από την πλευρά της Κομισιόν μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η διεύρυνση της Ευρωζώνης θα παραμείνει ανοιχτή, θα πρέπει να παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία. Εμείς από τη Σκοπιά της Κομισιόν καλωσορίζουμε τις χώρες που εργάζονται για την ένταξη στο ευρώ και είμαστε έτοιμοι να τις υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζεντιλόνι. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρεις ε, παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η εξής. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον, να περιορίζουμε κινδύνους και να συντονίζουμε τις δημοσιονομικές μας πολιτικές, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε 27 διαφορετικές δημοσιονομικές πολιτικές αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το γεγονός ότι χωρίς ε, ε, βαρότερο συντονισμό, να πω ε, ήδη έχουμε επιτύχει πολλά στο συντονισμό των πολιτικών μας, αλλά χωρίς ισχυρότερο συντονισμό δεν μπορούμε να αφήσουμε την οικονομική πολιτική μόνη της σε περίπτωση που προκύψουν πιο περίπλοκες καταστάσεις. Δεύτερον, με ρωτήσατε για τον ESM. Ναι, υπάρχει ε, γενική συμφωνία, αλλά οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Όσον αφορά λεπτομέρειες ή δευτερεύουσες πτυχές και αυτές οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και αυτή την επόμενη περίοδο υπό την ε, προεδρία του Μάριο Σεντένο στο Eurogroup. Τρίτη και τελευταία παρατήρηση. Ναι, έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά πολλές επιλογές. Ας πούμε όταν ακούω το γεγονός ότι η πρόοδος είναι πολύ αργή στην ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης αυτό εν μέρει οφείλεται ε, σε δυσκολίες στη διαδικασία αλλά για να μιλήσουμε ανοιχτά, αυτό κυρίως οφείλεται στις πολιτικές διαφορές. Οι πολιτικές διαφορές υπάρχουν και για το θέμα της ε, οικονομικής αναθεώρησης. Οι πολιτικές διαφορές λοιπόν υπάρχουν. Πώς μπορούμε να αναμίξουμε με πιο απλό αλλά ευέλικτο τρόπο και λύσεις όπως εσείς ζητάτε όλα αυτά δεν είναι καθόλου εύκολο. Το μόνο μου μήνυμα κυρίως προς τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι ότι για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες οι ευρωπαϊκοί θεσμοί χρειάζονται την πολιτική προσήλωση πίεσης και συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων σε αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει τεχνική λύση για αυτά τα προβλήματα χωρίς πολιτική βούληση. Και γι' αυτό είναι και ιδιαίτερα ευπρόζεκτη αυτή η κοινοβουλευτική εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Φάβιο Πανέτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συζήτηση. Νομίζω πως ε, ακούστηκαν πολλά ενδιαφέροντα σχόλια. Ε, δεν θα σχολιάσω με μονομένα κάθε ερώτηση, αλλά θα υπογραμμίσω κάποια ζητήματα που προέκυψαν. Αρκετά σχόλια εστίασαν στην ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Κεφαλαγορών και τη Τραπεζική Ένωση. Συμφωνώ απολύτω. Είναι ουσιαστικό στοιχείο αυτό για εμβάθυνση τη Νομισματική Ένωση, να βελτιωθεί ο ανταγωνισμό στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, να υπάρχει αμοιβοποίηση του κινδύνου ανάμεσα στου διάφορου επενδυτέ στα κρατημέλη και να βελτιώσουμε τι δημοσιονομικέ συνθήκες για την πραγματική οικονομία και αυτό αναφέρθηκε από αρκετούς ε, ομιλητές. Επίσης αναφέρθηκε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ενιαία αγορά και βέβαια όπως είπαμε η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαγορών θα μπορούσε να δώσει πρόσβαση σε διάφορες χώρες σε πλέον κεφάλαια. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε περαιτέρω προσπάθειες για να ολοκληρώσουμε αυτές τις δύο ενώσεις. Είναι όμως σημαντικό και για τη βασική εργασία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη εμβάθυνση τη Τραπεζική Ένωσης και το της των Κεφαλαγορών, αυτό θα σημαίνει ότι θα μας περιχαρακώσει από ε, δημοσιονομικά προβλήματα και σοκ και, αλλά θα βελτιώσει και τις δυνατότητες να μοιραστούμε ε, τα σοκ και άρα να έχουμε καλύτερο περιβάλλον για την εφαρμογή νομισματικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζών. Τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί πρόοδος γιατί έχει υπάρξει κίνηση πιο πιο προβλέψιμη και πιο διαφανή τραπεζική εποπτεία και αυτή είναι πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη. ασφάλεια τώρα και κυριαρχία των τραπεζών. Ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα είναι να βελτιώσουμε τη δημόσια οικονομία και πρέπει αυτό να το καταφέρουμε. Αναφερθήκατε στην ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες, οι δυνατότητες χρηματοδότησης, ειδικά στις μικρές εταιρείες. Ε, αν δούμε το γράφημα για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την δυναμική των ε, χρηματοδοτικών δανείων προς τις μικρές εταιρείες, θα δείτε ότι από την αρχή των μη νομισματικών πολιτικών από την ΕΚΤ, το κόστος για τις μικρές εταιρείε έχει μειωθεί πάρα πολύ, ειδικά για τις μικρές. Βεβαίως, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική θα τα καταφέρει να φτάσει η ανάπτυξη σε υπερβολικά ψηλά σημεία. Ε, Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αυτό σημαίνει, ε, συμβαίνει λόγω της συσνής ανάπτυξης από τις μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Το ξέρουμε αυτό με βάση τις αναλύσεις μας, αλλά θα πρέπει να δούμε τη δυναμική των ε, της δανειοδότησης που είναι ε, αυξανόμενη, αλλά να δούμε αν η ΕΚΤ δεν είχε ξεκινήσει αυτά τα μέτρα, τότε η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη για τα Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φυσικά θα πρέπει αυτό να προστρεχθεί στην Ευρωζώνη. Αυτό οφείλεται κυρίω. Βέβαια, βελτιώνονται τα πράγματα. Καλύτερε οικονομικέ συνθήκε είχαμε τελευταία χρόνια. Τώρα έχει σταθεροποιηθεί η ανάπτυξη. Αλλά ξανακολουθεί να είναι λιγοστή. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση για τι τράπεζε στι περισσότερε χώρε βελτιώνεται. Και εκεί όπου εντοπίζονται αδυναμίε, θα πρέπει να καλύπτονται μέσω παρεμβάσεων για τις γενικές οικονομικές πολιτικές ώστε να κινητοποιηθεί ανάπτυξη και σε εθνικό επίπεδο. Αυτά και ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στην Κρουσδάνα Πέριτς για τις τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν. Η Κροατία επιθυμεί τη διεύρυνση ε, της Ευρωζώνης ως προς τη χώρα μας. Γι' αυτό θέλουμε να συμμεριστούμε αυτό το κομμάτι της κυριαρχίας, όπως και άλλα κράτη. Αυτό που δημιουργήσε μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι νέοι θεσμοί και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που αφορούν την εποπτεία και εξυγίανση των τραπεζών ε, στο ενωσιακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει επέκταση της διακυβέρνησης, της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Με την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αυτό το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση. και με ένα ενιαίο σύστημα εγγύησης καταθέσεων και πρόσθετα μέτρα μείωσης των κινδύνων. Στην Τραπεζική Ένωση η ευθύνη για την προστασία και εγγύηση των καταθέσεων θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο ενωσιακό και το ίδιο ισχύει και για το μηχανισμό backstop. Υποστήριξη, ασφάλεια, προστασία και ασφάλεια. Ε, μιλήσαμε και για τους κινδύνους του κρυπτονομίσματος. Όλες αυτές είναι ε, αιτίες για να λύσουμε όλους τους κινδύνους και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ολόκληρης της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα ήθελα τώρα να κλείσω την Ολομέλεια που είχε θέμα ε, διεύρυνση και εμβάθυνση της ε, διακυβέρνησης της ΩΝΕ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους. Λύεται η συνεδρίαση αυτή. Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση θα συνεχιστεί στην Επιτροπή ΕΚΟΝ με μια άλλη συνεδρίαση που θα αρχίσει σε 15 λεπτά για το Διεθνές ε, Φορολογικό Σύστημα και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. την